So, ladies and gentlemen, are we ready to begin our afternoon meeting? Να ξεκινήσουμε. ξεκινήσουμε, κύριε και κύριοι. Our next point in the agenda. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι μια ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Πίτερ Μέλβι από την οργάνωση ΕΣΠΟΝ που προωθεί την περιφερειακή διάσταση μέσω γνώσης, μεταφοράς γνώσεων και ε, εκμάθηση πολιτικών. Και έτσι λοιπόν η ΕΣΠΟΝ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρατηρήσεων για τη Χωρική Ανάπτυξη και Συνοχή, προβάλλει διάφορα σενάρια για το 2050 για να αναπτύξει μια μακροπρόθεσμη προοπτική για την περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι να συνδράμει και να βοηθήσει τους ε, πολιτικούς ηθήνοντες για να έχουν ένα όρομα για τις ε, πόλεις και τις περιφερειές της Ευρώπης. Θα συζητήσουμε λοιπόν σήμερα τα αποτελέσματα, τα πορίσματα του οργανισμού ΕΣΠΟΝ και της εργασίας του και θα δώσω το λόγο στον κύριο Μέλμπι για να κάνει την παρουσίασή του. Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, να θέσουμε ερωτήσεις. Ελπίζω δε ο κύριος Μέλμπι να είναι σε θέση να απαντήσει στα ερωτήματά μας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την Επιτροπή που μας προσκάλεσε να σας ενημερώσουμε για τα αρκετά ενδιαφέροντα αυτά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά αυτή τη ε, μελέτη. Θα ήθελα να πω επίσης ότι ήταν και πολύ δύσκολο ε, εξ αρχής ε, το project αυτό. Είναι δύσκολη αυτή η πρόκληση του να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε σενάριο τόσο μακροπρόθεσμα και να παρουσιάσουμε και ενδεχόμενα οράματα για την πολιτική. Ξέρω ότι οι επιτροπές σας ενδιαφέρονται σε ό,τι αφορά το στρατηγικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Το θέμα λοιπόν αυτό ενδεχομένω να σας ενδιαφέρει ιδιαίτερω. Αυτό ελπίζω τουλάχιστον και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να σας δώσω κάποιε βασικές έννοιες για τα βασικά πορίσματα. Καταρχάς, να σα πω δύο λόγια για το πώ ξεκινήσαμε. Ήταν ένα από τα προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΣΠΟΝ, το οποίο αποφασίστηκε και απαιτήθηκε από όλες τις χώρες που ήταν πίσω από το πρόγραμμα ΕΣΠΟΝ 2013. 31 χώρες, η Κροατία δεν ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε που διαμορφώθηκε το αίτημα αυτό. Αλλά το αίτημα αυτό μας ζήτησε να κοιτάξουμε προς το μέλλον, να δημιουργήσουμε κάποια σενάρια για το μέλλον, γιατί όλοι γνωρίζουμε τις προκλήσεις που αντιμετώπιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και πριν το προσφυγικό άλλωστε. Και ξέρουμε ότι πολλές από τις προκλήσεις αυτές ε, επηρεάζουν την ε, χωροταξία, τις ισορροπίες στην Ευρώπη και τη χωρική ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν επιχειρήσαμε να αναπτύξουμε μια μακροπρόθεσμη προοπτική. Να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο αναφορά για την ανάπτυξη που θα μπορούσε ιδανικά να χρησιμοποιηθεί και από τους πολιτικούς αλλά και από τους ε, ειδήμονες ε, στον εκάστοτε κλάδο. Και φυσικά, όταν γίνονται τέτοιες ε, μακροπρόθεσμες μελέτες θα πρέπει κανείς να είναι προετοιμασμένος για το ότι θα πρέπει να υπάρξει και κάποιο σχέδιο δράσης, κάποιες συστάσεις, κάποιες οδοί για τις πολιτικές αποφάσεις που θα λεφθούν. Και αυτό λοιπόν ήταν ένα στοιχείο της έκθεσης, κάποιες συστάσεις. Δημοσιεύσαμε λοιπόν την έκθεση και θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι η όλη ιδέα πίσω από τη μακροπρόθεσμη ιδέα αυτή του σχεδιασμού της επικράτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των κρατών μελών. Στις 26-27 Νοεμβρίου να σας ενημερώσω ότι θα γίνει ανεπίσημη υπουργική συνάντηση στο Λουξεμβούργο στα πλαίσια της Προεδρίας του Συμβουλίου και έχουμε λοιπόν διαπιστώσει ότι όλο και πιο πολλές χώρες ενδιαφέρονται για αυτό το δύσκολο βήμα του να δημιουργηθεί ένα όραμα. Το όραμα είναι πάντα πολύ πολιτικό κομμάτι. Προαπαιτεί πολύ διάλογο, πολύ σχεδιασμό, πολύ συμμετοχή. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι τα συμπεράσματα της συνάντησης του Λουξεμβούργου και κατά πόσον θα ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Το δικό μας όμως το έργο και στο σημείο αυτό θα ήθελα καταρχάς να σας πω ότι σκόπιμα επιλέξαμε μια κλασική στρατηγική μεθοδολογία σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό μας και προσπάθησα να σας το δείξω αυτό στη διαφάνεια αυτή. Πρώτο λοιπόν βήμα είναι καταρχάς να καταγραφεί η κατάσταση, τα δεδομένα. Να δημιουργηθεί λοιπόν ένα σενάριο βάσης. Ένα σενάριο το οποίο γνωρίζετε ήδη ουσιαστικά, ε, δεν αλλάζει τίποτα, το πολιτικό μείγμα παραμένει ως έχει και έτσι απλά εξελίσσεται. Αυτό αποτελεί και το σημείο αναφοράς για όλο το πρόγραμμα. Και έτσι λοιπόν στην περίπτωση αυτή αναπτύχθηκαν και δύο, τρία διαφορετικά χωρικά σενάρια. Να τονίσω ότι πρόκειται για χωρικά σενάρια γιατί αφορά αυτό τρία ενδεχόμενα σενάρια για το μέλλον που θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από τις επενδύσεις, από πολιτικό μείγμα, το πολιτικό αμάγαλγαμα, προκειμένου να δημιουργηθεί μια είδους δομή στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Και θα σας δώσω και κάποιες φωτογραφίες, ε, θα σας δείξω και κάποιες φωτογραφίες. Καταρχάς λοιπόν για την προώθηση των μητροπολιτικών περιοχών. Και έτσι λοιπόν στα πλαίσια του ΩΣΑ μιλάμε πολύ για τέτοιες ε, γεωγραφικές ε, ενότητες. Ε, μία εξ αυτών είχε ως σκοπό την προώθηση τέτοιων ενότητων και των πόλεων, ενώ η τελευταία αυτή εκδοχή αφορούσε την προώθηση μικρών κομμοπόλεων και επίσης μειονεκτούντων περιοχών. Βλέπετε λοιπόν ότι στο γράφημα δημιουργείται ένας χαρταετός. Αυτός ο χαρταετός λοιπόν αποτελεί το σημείο όπου εντάσσεται το όραμα. Τέλος, το πέμπτο βήμα στην μέθοδο αυτή είναι να δημιουργηθούν και η οδή. Όταν διαμορφωθεί το όραμα θα πρέπει να συνοδευτεί από κάποιες ε, πολιτικές αποφάσεις, από κάποια βήματα τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν προκειμένου να επιτευχθεί το όραμα αυτό. Αυτά εισαγωγικά για να ξέρετε τι θα, σε τι να θα φερθώ στις διαφάνειες. Ας περάσουμε λοιπόν στο τρία εδαφικά σενάρια τώρα. Καταρχάς το σενάριο βάσης. Να σας ενημερώσω λοιπόν και να σας πω δύο λόγια γι' αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ παρουσιάζουν το εξή. Αυτά έχουν προετοιμαστεί από μια διεθνή ομάδα στην οποία έχει ανατεθεί το έργο αυτό. ειδική στην οικονομετρία, στη μοντελοποίηση. Άρα το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι μόνο αλλά και περιλαμβάνει παράλληλα πολλά αποσυντικά ζητήματα. Αν λοιπόν το σενάριο βάσης, αν η Ευρώπη συνεχίσει να αναπτύσσεται με το πολιτικό μείγμα το σημερινό, το αποτέλεσμα είναι ότι το ΑΕΠ ανά έτος θα αυξηθεί κατά 1,89% κατά πάσα πιθανότητα. Κοιτώντας όμως τις περιφέρειες, διαπιστώνουμε ότι έχουμε 44 περιφέρειες με ανάπτυξη κάτω από 1% μέχρι το 2030. Αυτό δεν πρόκειται λοιπόν να βλένει τις ανισορροπίες. Δεν πρόκειται να δημιουργήσει σύγκληση το να παραμείνει η κατάσταση δηλαδή όσο έχει σήμερα. Το πρώτο από τα περιφερειακά λοιπόν σενάρια. Και εδώ ασφαλώς η άσκηση αυτή είναι θεωρητική. Υπάρχουν πολλές εικασίες που υποστηρίζουν το σενάριο, δεν έχω χρόνο να επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά τα βασικά στοιχεία είναι ότι λέμε το εξής. Προσπαθούμε να υπογραμμίσουμε τον τρόπο που υποστηρίζουμε την εδαφική ανάπτυξη της ε, πολιτικές αποφάσεις ε, και έτσι οι 76 μικροπολιτικές ε, περιοχές στις οποίες έχουμε ορίσει στην Ευρώπη είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας σε ό,τι αφορά δηλαδή τις υποδομές, τις επικοινωνίες, τα δίκτυα και σε ορισμένες περιπτώσεις ε, δημιουργούνται κάποιες συνεργασίες μεταξύ των μεγάλων πόλεων αυτών για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους στο παγκόσμιο προσκήνιο. Τέτοιου είδους λοιπόν σενάρια θα δείτε ότι έχουν και μια, ένα εδαφικό αποτύπωμα, το οποίο το βλέπετε στα αριστερά, στην ε, φωτογραφία. Αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά το μέλλον ε, της εδαφικής ε, διάστασης. Το επόμενο αφορά την πρόθεση των δικτύων πόλεων, ίσως το δεύτερο επίπεδο συνένωσης και συνεργασίας. Εδώ έχουμε 261 πόλεις και δημιουργεί ένα εδαφικό ίχνος. Όπως βλέπετε είναι λίγο πιο ισορροπημένο, φτάνει στις γωνιές της Ευρώπης, είναι πιο απλωμένο το δίκτυο αυτό ε, και στοχεύει στην ε, ισόρροπη ανάπτυξη. Τρίτο σενάριο που αφορά τις μικρότερες πόλεις και τις ε, περιοχές που έχουν μείνει λίγο πίσω σε ό,τι αφορά την ανάπτυξή τους. Και εδώ βλέπουμε ότι είναι ακόμα πιο απλωμένο. Ας δούμε λίγο τις διαφορές και ας συγκρίνουμε τα σενάρια. Έχουμε δύο ημερομηνίε στόχου, 2030 και 2050. Σε ό,τι αφορά το 2030, για το οποίο έχει και περισσότερο νόημα να κάνουμε μοντέλα, αν συγκρίνουμε τα τρία σενάρια, προκύπτει ότι το σενάριο που προωθεί τις μετροπολιτικές περιοχές και τις πόλεις, αυτά τα δύο σενάρια ε, δημιουργούν περίπου ίδια ανάπτυξη, δύο ανάπτυξη, ενώ το σενάριο Γ είναι λίγο πιο πίσω. Αν δείτε το εδαφικό ίχνος, θα δείτε το σενάριο Β είναι αυτό που δίνει το μεγαλύτερο επίπεδο ανταγωνιστικότητας και συνοχής. Αυτό που δεν φαίνεται στο χάρτη είναι ότι οι διαφορές μεταξύ των περιφερειών θα μειωθούν κατά πολύ λίγο μέχρι το 2030. Τώρα για το 2050 Δηλαδή, μακροπρόθεσμα, η οικονομική ανάπτυξη δεν θα επηρεαστεί οποιοδήποτε από τα τρία μοντέλα και αν επιλέξουμε. Αυτό αποδεικνύει ότι αυτό δίνει μεγάλο περιθώριο σε ό,τι αφορά την πολιτική που θα επιλεγεί γιατί κατά βάση όλα τα σενάρια αυτά είναι εφικτά, δεν θα πληγεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν επιλέξουμε για παράδειγμα ένα σενάριο το οποίο θα είναι πολύ πιο ισόρροπο και ισοκατανεμημένο. Αυτό είναι ένα από τα βασικά πορίσματα του έργου αυτού. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο αμφισβητείται, αν θέλετε, το αποτέλεσμα και διαφόρων μελετών, εντάξει αυτών και του ΟΣΑ, που, ε, που ε, θεωρούν πως η προώθηση των μητροπολιτικών περιοχών ε, έχει περισσότερα πλεονεκτήματα. Δεν είναι λάθος ότι έχει πλεονεκτήματα, αλλά δεν είναι και όλη η αλήθεια. Ακόμα και αν δεν προωθήσουμε τις μητροπολιτικές προοχέ τόσο πολύ, η ανάπτυξη στην Ευρώπη θα είναι περίπου ίδια. Και με αυτές τις διαφάνειες προσπαθούμε να σας δείξουμε και την εξέλιξη. χωρίς ε, να παρεμποδίσουμε την οικονομική ανάπτυξη μπορούμε να επιλέξουμε μια ανάπτυξη που θα πηγαίνει, ε, θα ακολουθεί αυτή την πορεία που βλέπετε εδώ 2020, 2030, 2050. Εδώ είμαστε πλέον στο 2050, όπου βλέπετε και την ε, ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ της Ευρώπης και των γειτονικών της χωρών. Όλα αυτά δημιουργούν την πλατφόρμα για το όραμά μας επί τη βάση των τριών σενάριων. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ένας τίτλος που λέει κάνοντας την Ευρώπη πιο ανοιχτή και πολυκεντρική. Ανοιχτή με στόχο να ενώσουμε την Ευρώπη με τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι ώστε η Ευρώπη να μην μείνει πίσω, να εξακολουθεί να είναι ατμομηχανή της παγκόσμιας ανάπτυξης. Ε, επίσης, προώθηση της ε, συνεργασίας με τις γειτονικές περιοχές και την παράλληλη, την πρόθεση παράλληλης ανάπτυξης. Πολυκεντρική Ευρώπη ε, είναι προφανές τι είναι αυτό, αλλά είναι επίσης και μια πιο ισορροπημένη αστική δομή με αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής ανάπτυξης ε, πάνω στις, ε, στους πόρους. Σε κάθε ένα από, τους, από αυτούς τους στόχους ε, έχουμε και κάποια πιο λεπτομερή πράγματα. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο να σας τους παρουσιάσω. Ίσως ενδεχομένως ό,τι αφορά το πρώτο, την παγκόσμια, την, την ένωση της Ευρώπης με τον υπόλοιπο κόσμο, ε, αυτό σημαίνει άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών, βελτίωση της ε, αποτελεσματικότητας σε ό,τι αφορά τις συνδέσεις, έτσι ώστε πρόσωπα και εμπορεύματα μπορούν να μεταφερθούν εύκολα, καθώς επίσης και η, η δημιουργία του Διευρωπαϊκού Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ευρωπαϊκού Ηλεκτρικού Δικτύου ε, κλπ. Ε, όταν μιλάμε για ε, ισορροπημένη δομή, μιλάμε για την πρόθεση ε, πιο μεσαίων περιοχών και περιφερειών και πόλεων ως ατμομηχανές της ανάπτυξης. Ε, ε, όπου θα ε, αναπτύσσονται όλες οι, όλα τους τα τμήματα και βέβαια ε, ένταξη των λειτουργικών αστικών περιοχών. Ε, μην ξεχνάμε ότι το μεταναστευτικό ή το προσφυγικό θα δημιουργήσει αλλαγές, θα προκαλέσει αλλαγές και θα δημιουργηθούν πολλές καινούριες ανάγκες και καινούριες προτιμήσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη στο, στην ανάλυση που κάνουμε για την περίοδο μέχρι το 2030-2050. Στην τελευταία διαφάνεια θέλω να σας δείξω πώς μπορούμε να παρουσιάσουμε το εδαφικό μέλλον της Ευρώπης αυτή τη στιγμή αριστερά βλέπετε το αποτέλεσμα ε, της ε, παράλληλης των διαφόρων δράσεων ε, και πολιετών σχεδίων. Αν όμως επιβεβαιωθεί μια πολιτική βούληση να προχωρήσει σε κάτι πιο ευρωπαϊκό, τότε η εικόνα θα πρέπει να είναι αυτή του δεξιού κομματιού. Ε, όχι ακριβώς ενδεχομένω διότι όλα θα εξαρτηθούν από τι ακριβείς πολιτικές επιλογές, αλλά ο χάρτη θα πρέπει να έχει αυτή τη μορφή. Ε, αυτό το μοντέλο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για μια σειρά πολιτικών. Αυτά εισαγωγικά έχω τρία έγγραφα μαζί μου. Το ένα από αυτά είναι το έγγραφο κλειδί, το βασικό έγγραφο που παρουσιάζει τα, βασι... κύρια στοιχεία και τα επιχειρήματα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη ενό τέτοιου οράματο, εδαφικού οράματο. Και μετά έχουμε και άλλα δύο έγγραφα, αυτό που είναι στο κέντρο και αυτό που είναι δεξιά, που αφορούν πιο πολύ αυτούς που θέλουν να μάθουν λίγο περισσότερα, λίγα περισσότερα πράγματα για τις παραδοχές πίσω από τα διαφορά. Τα τρία δηλαδή σενάρια. Ίσως δεν έχουμε αντίγραφα για όλους, αλλά έχουμε αντίγραφα εδώ στην αίθουσα και αν θέλετε μπορείτε να τα δείτε και να τα πάρετε. Αυτά εισαγωγικά ελπίζω να σας ε, ενέπνευσα ενδιαφέρον. Από ό,τι φαίνεται όλα αυτά έχουν ήδη εμπνεύσει τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος, για την παρουσίαση. Έχουμε, θέλω να ελπίζω πράγματι, αντίγραφα για όλους, <clears throat> για όλα τα μέλη της Επιτροπής. Αν δεν έχουμε, θα φροντίσουμε να αποκτήσουμε. Συνάδελφοι, έχετε το λόγο για ερωτήσεις, σχόλια κτλ. Ο κύριος Βανίστερο Ευχαριστώ για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση που μας είπατε την αρχή ότι θα ήταν ενδιαφέρουσα σχετικά με τις δυνατότητες που έχουμε να κάνουμε συγκεκριμένες επιλογές όχι μόνο για μία κατηγορία του εδάφους, τις πιαστικές περιοχές ή τις λιγότερο και προκειμένου να μην έχουμε έντονα διαφοροποιημένες καταστάσεις στο ευρωαϊκό, στην ευρωαϊκή εδαφική πραγματικότητα το οποίο εκπλήσει γιατί ε, κανείς σκέπτεται πάντα ότι οι μητροπολιτικές αστικές περιοχέ είναι αυτές που πάντα ηγούνται και θα ηγούνται και στο μέλλον εάν κάτι τέτοιο δεν αν δεν προκύπτει ότι μόνο πολλούν την κατεύθυνση δεν ξέρω τι μπορούμε να αλλάξουμε στην Ευρώπη ακόμα και όταν έχουμε επιστολές ας πούμε από τον Πρωθυπουργό Κάμερον. Εν πάση είδαμε τα τελευταία χρόνια της κρίσεως μια ισότιμη μάλλον ότι αυτά τα χρόνια της κρίσεως δεν είναι δεν εξισορροπήθηκαν οι μορφές στήριξης προς τις, δύο, προς τις διάφορες εμπάσχερτός ιδαυκές πραγματικότητες Ευρώπης μεταξύ των αστυνικών και της υπαίθρου δηλαδή εννοώ. If to our general aims in the cohesion... Αν δω τους γενικότερους στόχους της πολιτικής μας συνοχής και εν ώψη της ε, κατεύθυνσης της παγκόσμιας και παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, τι θα λέγατε, πώς θα λέγατε ότι θα μπορούσαμε να επιλύσουμε αυτήν την ε, έλλειψη ισόρροπης αντιμετώπισης. Και από ό,τι ακούμε από τις συναντήσεις του Συμβουλίου υπάρχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για, τα, για τις εδαφικές ε, πτυχές να εξετάσουμε κάτι τέτοιο και να το συσχετίσουμε με τις μεταφορές, με όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Οπότε η ερώτησή μου, λέει ο κ. είναι πού πιστεύετε ότι θεωρείτε ότι λαμβάνεται υπόψη, λαμβάνεται με αλφαγιώτα υπόψη αυτό το στοιχείο και πώς διαχέεται. Δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να συναντήσουμε και να συζητήσουμε με ανθρώπους που είναι ενημερωμένοι σχετικά με αυτά που μας παρουσιάσατε. Πώς επικοινωνείτε εσείς με τους πολιτικούς ηθήνοντες κρατών, πόλεων και ενώσεως. Ευχαριστούμε κύριο Σόλμπρεχτ. <coughs> this is very ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση αυτή και νομίζω ότι πρέπει να την εξετάσει κανείς ε, προσεκτικά. Και συνάδει και με την συζήτηση για, την, για το μέλλον τη ε, πολιτική συνοχής. Και νομίζω ότι ακούσαμε και τα τρία σενάρια για τις μεγααστικές περιοχές, τις αστικές περιοχές και τις υπόλοιπες περιφέρειες γιατί σε όλα τα σενάρια πράγματι υπογραμμίζεται ο ρόλος των αστικών περιοχών. Γιατί ακόμα και για τις υπόλοιπες περιφερειές αναφερόμαστε σε πόλεις μεσαίας κλίμακας. Επομένως, μήπως θα έπρεπε κανείς να συμπεράνει ότι η περιφερειακή πολιτική, είτε το θέλει κανείς είτε δεν όχι, είτε όχι, είναι πολύ πιο εστιασμένη στην αναπτυξιακή πολιτική των πόλεων, όλων των ιδίων των πόλεων, από τις Μητροπόλεις μέχρι τις Κομοπόλεις. Γιατί αν αυτό είναι αλήθεια σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που επαναλαμβάνουμε συνεχώς, δηλαδή την αστική πολιτική. Εκτός αν υπεραπλωστεύω, γιατί αυτό κυρίως εννοούμε με την περιφερειακή πολιτική στην ουσία. Επίσης για τα ΝΑΤΣ, 1, 2, 3 κτλ. Έχουμε το βασικό επίπεδο της καταχώρησης των περιφερειών επί τη βάση του ΝΑΤΣ 2 και του ΑΕΠ ως μοναδικά κριτήρια. Όταν βλέπω τα τρία σενάρια συμπεραίνω ότι μάλλον το πιο ρεαλιστικό είναι το δεύτερο σενάριο που βασίζεται στο ΝΑΤΣ 2 και το ΝΑΤΣ 3 είναι ενδιαφέρον αλλά το πιο ενδιαφέρον για το μέλλον λέει ο μιλτής είναι το ΝΑΤΣ 2 Επομένως, το επίπεδο από ό,τι φαίνεται για το μέλλον το καταλληλότερο είναι το ΝΑΤΣ 2. Ε, ή, μήπως θα έπρεπε να κινηθεί κανείς προς το ΝΑΤΣ 3 και 4. Πώς βλέπετε τις κατευθύνσεις της Κομισιόν. Πώς μπορεί να μεταφραστεί δηλαδή η εδαφική συνοχή σε μια πιο απτή πολιτική. Γιατί από το υλικό αυτό που μας δείξατε φαίνεται ότι το ΝΑΤΣ 2 δεν είναι ότι συνεχίζουμε ως συνήθως και ότι ίσως θα ήταν το καταλληλότερο, καταλληλότερη προσέγγιση. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, για την περιφερειακή πολιτική, αυτά. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, η κυρία Μπρέσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέει η κυρία Μπρέσο. Μία παρατήρηση και μία ερώτηση. Ε, στο πλαίσιο της προώθησης των πόλεων που αναφέρθηκαν και οι συνάδελφοι, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μία μονοεστίαση ε, σε πρωτεύουσες, σε αυτό το μικρό γράφημα που είναι δύσκολο να το δει κανείς, αλλά εστίαση που ίσως να αντιστοιχεί σε μια χώρα σαν τη Γαλλία, αλλά όχι σε μια δομή αντίστοιχη με την τωρινή και μελλοντική της δικής μου της χώρας. Γιατί με όλα τα μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης που έχουμε στην Ιταλία, με μερική εξαίρεση ενδεχομένως της δικής μου περιφέρειας του Πιεμότε, έχουμε αναπτυχθεί από το Μιλάνο και προς τα έξω. Από το Μιλάνο προς τα έξω. Και χωρίς να φτάνουμε αναγκαστικά μέχρι τη Ρώμη το οποίο ίσως να μην αντιστοιχεί ούτε στο παρελθόν και ούτε και στο μέλλον. Δηλαδή σε αντίθεση με το γαλλικό μοντέλο που σας περιγράφω η Ιταλία είναι πολυκεντρική χώρα και ίσως αυτό να ισχύει και για άλλες χώρες. Ίσως. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα μοντέλο που βασίζεται στις πρωτεύουσες και μέσω της πολιτικής συνοχής ενισχύεται ο ρόλος της πρωτεύουσας. και δημιουργεί εσωτερικές δυναμικές διαφοράς, διαφοροποίησης εντός της χώρας. Γιατί υποτίθεται ότι η γενική μας στόχη είναι η σύγκληση της οικονομίας και όχι η απόκληση και μπορεί να επιτυγχάνουμε, αν την επιτυγχάνουμε, τη σύγκληση σε επίπεδο αλλά όχι στο ιστορικό των χωρών, όπου κάνουμε το αντίστροφο. Τώρα, ναι, οκ, okay, προώθηση των πόλεων, των αστικών κέντρων, αλλά ή στα πλαίσια ενό αποκεντρωμένου και πολυκεντρικού, εν πάση περιπτώσει, συστήματος. Και όχι μόνο επί τη βάση της πρωτεύουσα. Πρώτον, αυτό. Δεύτερον, στην Ευρώπη αναπτύσσεται αρκετά δυναμικά η στρατηγική, η μακροπεριφερειακή, η οποία αναφέρεται σε μία εδαφική αναδιοργάνωση της Ευρώπης που βασίζεται σε μία αρχή περισσότερο bottom-up. Δηλαδή επιλέγονται αν θέλετε οι συγκεκριμένες περιοχές που είναι περιοχές ανάπτυξης. η εδαφική αρχή που έχει εγγραφεί στη Λισαβόνα οθεί και εξωθεί προς μια μεγαλύτερη διασυνοριακή συνεργασία ή στα πλαίσια μιας λογικής που έχει σχέση με το έδαφος, έχει σχέση με τις ιστορικές παραδόσεις, τις οικονομικούς πόρους, τη γεωγραφία, τα όρη, της υδάτινες οδούς αλλά οπωσδήποτε υπάρχει μια ιστορική και παραδοσιακή δομή που μετατρέπεται, μεταφράζεται σε απτές και συγκεκριμένες στρατηγικές. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να διατηρείται υπόψη σε οποιαδήποτε στρατηγική ανάλυση, διότι αν θέλετε διαφοροποιείται αυτή τη στιγμή η εδαφική και γεωγραφική διάσταση της οικονομικής συνεργασίας και της ανάπτυξης. Ευχαριστούμε, λέει η πρόεδρος, η κυρία Βάνα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση, η οποία πραγματικά ήταν εξαιρετική. εξαιρετική. Και για την ε, παρουσίαση. Ήθελα να ρωτήσω για την μέθοδο και για τους δείκτες που, που χρησιμοποιήσετε. Χρησιμοποιείτε ως βασικό δείκτη για την κοινωνικονομική ε, ανάπτυξη το ΑΕΠ ως ήθιστη ή προχωράτε λίγο τις ε, έννοιες αυτές της κοινωνικο-οικονομικής εξέλιξης και ανάπτυξης, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάποιες περιπτώσεις, σε ό,τι αφορά δηλαδή την ε, περιφερική ανάπτυξη, θέματα φτώχειας, ε, περιβάλλοντος, εκπαίδευσης, παιδείας, για να δημιουργήσετε μια πιο ευρεία διάσταση. Νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο μια υπηρεσία όπως η ΕΣΠΟΝ να δημιουργήσει μια τέτοια ευρεία διάσταση στην ε, ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο Πρόεδρος, ε, καμία άλλη ερώτηση. Θα ήθελα και εγώ ως μέλος ε, της Επιτροπής Ρέτζη να θέσω μια ερώτηση. Θα μιλήσω στη γλώσσα μου, στα βουλγαρικά. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό η προοπτική περιφερειακής ανάπτυξης ε, της Ευρώπης, ε, όπως την παρουσιάσατε στην Ευρώπη, ανταποκρίνεται στην ε, προγραμματική περίοδο 2014-2020. Πιστεύετε ότι τα σενάρια τα οποία μας αναφέρατε καταρτίστηκαν όταν ε, υπογράφτηκαν οι σχετικές συμφωνίες ε, εταιρικές σχέσεις και τα σχετικά προγράμματα. Και αυτό το ρωτώ, μιας και προερχόμαι από μια χώρα, μιας και εκπροσωπώ μια χώρα η οποία προσπαθεί να διατηρήσει μια ανάπτυξη σε πολλαπλά, με πολλαπλά κέντρα. Παρ' όλα αυτά, οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής μας πρόχνουν ουσιαστικά προς ένα μοντέλο κάθε άλλο παρά το οποίο θα συνεπαγόταν ότι θα υπήρχαν δύο-τρία κέντρα ανά χώρα, αλλά ότι θα αγνοούσαμε ουσιαστικά τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που υπάρχουν σε άλλες πόλεις, σε πιο μικρές πόλεις, σε πιο μικρά κέντρα, τα οποία είναι σημαντικά για τις περιφέρειες, αλλά όχι απαραίτητα σε σημείο προτεραιότητά για την πολιτική συνοχή που εγκρίνεται και εφαρμόζεται. Αν συνεχίσουμε λοιπόν να συζητάμε αυτά τα σενάρια, αυτές τις εικασίες, τι θα γίνει την περίοδο μετά το 2020, πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε ένα πακέτο για την ε, πολιτική συνοχή προκειμένου τα κράτη-μέλη να έχουν την επιλογή φυσικά ανάλογα και με τι ε, πολιτικές τους επιλογές στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να υπάρχουν πολλοί κέντρες, αν θέλετε, τα μοντέλα ανάπτυξη και όχι μόνο ομόκεντρο. ανάπτυξη. Τελευταία ερώτηση ήταν αυτή, λέει η Πρόεδρος. Δεν βλέπω κανέναν άλλον να ζητάει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, συγγνώμη που ζητώ το λόγο μετά από σας, αλλά με ενέπνευσε η ερώτησή σας. Ε, θέλω να δώσω το παράδειγμα της Πορτογαλίας. Η διαφορά ανάμεσα στις περιφέρειες έχει σχέση ε, όχι μόνο με πολυκέντρισμα, πολλές φορές και με πόλωση. Ε, οι χώρες που ακολούθησαν τον πολυκεντρισμό νομίζω ότι εξεφάλισαν μεγαλύτερη αρμονία στην ανάπτυξή τους. Στις ε, περιφέρειες στις οποίες επικράτησε πόλωση, ε, η ανάπτυξη ανακόπηκε. Οπότε το μοντέλο της πολυκεντρικής ανάπτυξης που έχει προφανώς τεράστια πλεονεκτήματα δεν θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα. Ή εν δεν είναι το μοντέλο πιο πολύ ωφελεί την ανάπτυξη έναντι ενός μοντέλου πόλωσης. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Ε, ξέχασα να πω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιπροσωπεύεται. Ο κ. Φιλίπ Μονφόγ είναι μαζί μαζί μας Έχω δίκιο. Θέλετε να πάρετε το λόγο κύριε Μονφόρ τώρα ή αργότερα μετά τις απαντήσεις. Να πω δύο λόγια τώρα. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω. Θέλω μόνο να πω ότι το ε, έργο αυτό είναι σημαντικό μέσα στο πρόγραμμα ΕΣΠΟΝ. Είναι μια ανάλυση που αφορά πολλά, τα, ε, πολλά μελλοντικά χρόνια. Οι μέθοδοι και οι δείκτες που χρησιμοποιούμε συζητήθηκαν πάρα πολύ ε, και είναι πολύ σημαντική για, αυτή την, για τέτοιου αναλύσεις. Το σημαντικό μας για αυτό το project είναι ότι ε, παρόμοι, όπως και, με, και άλλες αναλύσεις συμφωνεί στο ότι το, ο μηχανισμός σύγκλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ακόμα και αν δεν έχει διαλυθεί και καταστραφεί έχει ε, χάσει δυναμισμό και η σύγκληση καθυστερεί. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για να προχωρήσουμε στο μέτωπο της σύγκλησης και να πετύχουμε μια ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα δεδομένου ότι αντιμετωπίζουμε σημαντικές καινούριες προκλήσεις, σε οποίες αναφέρθηκε και ο Πίτερ. Προκλήσεις και εντός και εκτός των συνόρων μας. Κομισιόν πιστεύει ότι τέτοιου είδους ανάλυση του, αναλύσεις του για το μέλλον είναι πολύ σημαντικές για να δούμε λίγο μπροστά και να αποφασίσουμε πώς θα σχεδιάσουμε τα προγράμματα και τις παρεμβάσεις μας στο μέλλον. Οπότε στηρίζουμε τέτοιου είδους αναλύσεις και προφανώς ε, συμμετέχουμε. Ωραία. Κύριε Μέλμπη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ για τα επενετικά σχόλια. Να πω και σας κύριε Πρέτσι ότι δεν πρόκειται για πρωτεύουσες και μητροπολιτικές περιοχές. Τα βασικά αποτελέσματα είναι, το βασικό αποτελέσμα είναι ότι δεν χρειάζεται να πιστέψουμε ε, τόσο πολύ όσο στο παρελθόν ότι μόνο μετροπολιτικές περιοχές μπορούν να αποτελέσουν ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας. Υπάρχουν και πόλεις δευτέρου επίπεδου με πολύ δυναμικό, με πολλές δυνατότητες ανάπτυξης, το είδαμε και πριν την κρίση και το οικονομετρικό μοντέλο πίσω από αυτήν την ανάλυση δείχνει ότι ο δείκτη ανάπτυξη, για τα επόμενα 15 χρόνια θα είναι περίπου ίδιος είτε ακολουθήσουμε το πρώτο μοντέλο είτε ακολουθήσουμε το δεύτερο. Αυτό είναι το βασικό ε, συμπέρασμα, ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε και ένα πολυκεντρικό μοντέλο. Ίσως στην πρώτη φάση μέχρι το 2030 θα πρέπει μάλιστα να ενθαρρύνουμε και να προωθήσουμε την ανάπτυξη των ε, πόλεων δευτέρου επίπεδου. Αυτό σίγουρα θα δημιουργήσει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης στην Ευρώπη με το αν ακολουθούσαμε το μοντέλο το μητροπολιτικό. Και ίσως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και την περαιτέρω ακόμα διεύρυνση των επενδύσεων, εδαφικά εννοώ. Αυτά θα τα δείτε εσείς ως πολιτικοί, εσείς μαζί με άλλους πολιτικούς. Εσείς θα πρέπει να καθορίσετε ένα πλαίσιο αναφοράς με την στήριξη των κρατών μελών, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα είναι ε, υποχρεωτικής εφαρμογής, ε, ότι δεν θα είναι δεσμευτικό, το συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια. Νομίζω ότι ένα πλαίσιο αναφοράς θα ήταν καλό και χρήσιμο και θα είχε και θετική επίπτωση, θετικές συνέπειες πάνω στην ε, ε, στο σχεδιασμό πολιτικής. Οπότε θα μπορούσαμε να πάρουμε οποιοδήποτε αυτά σενάρια και να τα αναμίξουμε κιόλα. Ε, ή να ακολουθήσουμε το ένα μετά το άλλο για διαφορετικές χρονικές περιόδους. Εσείς θα τα δείτε όλα αυτά, εσείς θα τα συζητήσετε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πώς θα πλησιάσουμε τον κόσμο και πώς θα επηρεάσουμε ευρύτερες μάζες νομίζω ότι θα φτάσει στους υπουργού 26 και 27 του μηνός εκεί θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε τα μάτια και των υπουργών που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, για την περιφερειακή ανάπτυξη και τα εδαφικά ζητήματα Οι υπουργοί λοιπόν θα ενημερωθούν στο τέλος του μήνα. Σίγουρα όμως πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Χρειαζόμαστε πιο πολύ διάλογο, χρειαζόμαστε ε, προκαταβολικά να ε, προωθήσουμε τα συμπεράσματα, να τα διαδώσουμε και να πείσουμε. Νομίζω ότι ο στόχος δεν είναι να τα συγκεντρώσουμε όλα στο κέντρο της Ευρώπης. Αυτό από πολιτικής πλευράς δεν είναι αποδεκτό όραμα. Το όραμα της Ευρώπης είναι μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη και πιο πολυκεντρική δομή. Το project αυτό εστίασε βέβαια περισσότερο στις πόλεις, αλλά όχι μόνο στις πρωτεύουσε. Πολλές πόλεις σε κάθε χώρα και βέβαια ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες χώρες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. στην Ευρώπη υπάρχουν περιοχές για τις οποίες χρειάζονται ιδιαίτερες προσπάθειες παρέμβασης, χρηματοδότησης, ε, ε, απειλούνται από την αστιφιλία, από τις αλλαγές του κλίματος κλπ. Από την άλλη μεριά θα πρέπει οι πόλεις πια να είναι λειτουργικές σε ένα πολύ ευρύτερο περιβάλλον έτσι ώστε η κατάσταση να είναι προς αμοιβαίο όφελος όλων. Η, ο πιο δύναμος κρίκος είναι ύπεθρος, αλλά θα πρέπει να βοηθηθεί να αναπτυχθεί, όχι να παρεμποδιστεί από τις πόλεις. Ε, οι, μα, οι στρατηγικές, μακροπεριφερειακές στρατηγικές προφανώς είναι τμήμα, το λέμε στην ε, έρευνά μας, στη μελέτη μας, ε, προωθούν την ε, διασυνοριακή ανάπτυξη. Οι μακροπροσιακές ε, στρατηγικές είναι ένα στοιχείο διασυνοριακής συνεργασίας. Στο άλλο άκρο ακόμα και τα όρια μεταξύ κοινοτικών διαμερισμάτων υπάρχουν ως σύνορα. Μερικές φορές και εκεί πρέπει να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία διότι θα δημιουργηθούν πλεονεκτήματα από, την, ε, από τον άλληλο ερεθισμό, από την συνεργασία και την, και την ανάπτυξη. Ε, παρουσιάζουμε συγκεκριμένους δείκτες για το ΑΕΠ, ε, παρουσιάζουμε συγγνώμη το ΑΕΠ ως συγκεκριμένο δείκτη, αλλά υπάρχουν και άλλοι δείκτες στους οποίους συμπεριλάβαμε στο σενάριο. Κοιτάξτε το υλικό και θα δείτε και τους υπόλοιπους δείκτες που χρησιμοποιήσαμε. Δεν είναι δυνατόν προφανώς να στηριχθούμε μόνο σε έναν δείκτη. Το μοντέλο που χρησιμοποίησαμε δεν είναι μόνο οικονομετρικό, ε, είναι και μεταφορικό και νομίζω και περιβαλλοντικό σε κάποιο βαθμό. Τέλος, για την ερώτηση Προέδρου, αν ε, μιλάμε για την πολιτική συνοχή μετά το 2020, τότε όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο. Αν μπορούσαμε να διαθέτουμε ένα πλαίσιο αναφορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για το ποιο είναι το όραμά μας για την πολιτική συνοχή μετά το 2020, αν όλα αυτά μπορούσαμε να τα εντάξουμε στη σκέψη μας, αυτό θα ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμο. Και ίσως έτσι θα μπορούσαμε να κατευθύνουμε κατά κάποιο τρόπο και τις επενδύσεις και τις προτεραιότητες της επόμενης φάσης της πολιτικής συνοχής. Ίσως βέβαια είναι λίγο απατηλά όνειρα, φρούδες ελπίδες, αλλά θα ήταν χρήσιμο. Η παγκόσμια κατάσταση είναι πολύ ρευστή, η Ευρώπη μένει πίσω, άλλες ε, ήπειροι διαμορφώνουν τέτοιου είδους στρατηγικές ήδη, οπότε ίσως είναι η στιγμή και για την Ευρώπη να ξεκινήσει κάτι αντίστοιχο. Σε ό,τι αφορά τις ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης, ε, ε, σίγουρα το project αυτό δεν τις επηρέασε, ε, ήρθε πολύ καθυστερημένα, ίσως μια επόμενη φορά. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και για, ευχαριστώ και για την ανταλλαγή απόψεων. Σε ευχαριστώ κύριε Σφαλίσσεράη. Να σχολιάσω για το θέμα που έθεσε ο Γιάνν Ολμπρέιχτ για τον ΑΤΣ 2, για τον σχεδιασμό. Και επίση για την παρατήρηση για τα σενάρια. σε ό,τι αφορά την περιφερειακή πολιτική και τη συμπερίληψη των πόλεων αυτών. Αυτό ενδεχομένως να μην είναι τόσο περίεργο να συνεχιστεί. Να δύο λοιπόν το πεδίο ε, λειτουργίας και η περιφερειακή πολιτική να συμπεριλάβει και τις πόλεις ως μοντέλο ανάπτυξης. Θα μπορούσατε να τα σχολιάσετε αυτά. Κοιτάξτε, δεν θέλω να πω πολλά για το ΝΑΤΣ 2. Θα ξέρετε κι εσείς ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ της ε, φυσικής περιφέρειας η οποία ορίζεται ως ΝΑΤΣ 2 από χώρα σε χώρα. Είναι κάπως επικίνδυνο να δηλώσουμε ότι κάνουμε σχεδιασμό βάσει των περιφερειών ΝΑΤΣ 2. Θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με την πραγματικότητα στο μέλλον. Αυτή η έννοια των ε, λειτουργικών περιφερειών ορισμός στο σωστό επίπεδο προκειμένου να ληφθούν οι σωστέ αποφάσεις, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όσο πιο μεγάλο δυναμικό γίνεται. Δεν θα ήθελα απαραίτητα να κάνω τη σύνδεση με μια πολυτεχνική ονοματολογία. Φυσικά αναγκαζόμαστε στις στατιστικές να χρησιμοποιήσουμε τέτοια δεδομένα, τέτοιες ποσοτικές πληροφορίες. Και αυτό το ίχνος ενδεχομένω να το βλέπετε, να το διακρίνετε. Αλλά δεν πιστεύω ότι στην πραγματικότητα θα πρέπει να αισθανόμαστε περιορισμένοι στο πώς ε, ορίζουμε τις ε, περιοχές σχεδιασμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις πόλεις. Νομίζω ότι σωστό είναι να ληφθεί ως βασικός παράγοντας το αστικό στοιχείο για τη διαμορφώση των εκάστοτε σενάριων. Αλλά σας είπα ότι είναι και σημαντικό να μην ε, παρακάμψουμε, να μην αγνοήσουμε την πραγματικότητα η οποία δεν είναι τόσο ρόδινη σε πολλά τμήματα της Ευρώπης. σε ό,τι αφορά και τις παρεμβάσεις στην πολιτική στο πλαίσιο αναφοράς, στο τι θέλουμε δηλαδή να πετύχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και ένα σενάριο το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και τις προκλήσεις της υπέτρου. Αλλά και τις ε, περιοχές υπέτρου που είναι κοντά στις πόλεις, κοντά σε αστικά κέντρα και αυτές λοιπόν θα πρέπει να ενταχθούν στα σχέδια προκειμένου να υπάρχει ένα θετικό μέλλον για τις περιοχές αυτές στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίο σχόλιο του κυρίου Άλμπρεχτ. Ζητώ συγγνώμη που επανέρχομαι. Ένα σύντομο σχόλιο. Καλό είναι να λέμε ότι εξαρτάται από τους πολιτικούς ηθήνοντες. Καλό και ευφυέ. Το θέμα είναι ποιο θα αναλάβει την ευθύνη. Αλλά το ΝΑΤΣ δεν είναι μόνο στατιστικά δεδομένα. Είναι κρίσιμη σημασία για τη λήψη αποφάσεων στην πολιτική. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον στο σύνολο της διαδικασίας. Όταν μιλάτε για τη συνάθρηση, των ΝΑΤΣ 2 κτλ. Διατηρούμε στην, στην πραγματικότητα την πολιτική όσο έχει σήμερα. Αν, ε, αν θέλουμε όμως να διαμορφώσουμε την πολιτική προς τις συνθήκες, Χρειαζόμαστε διαφορετικά νατς για διαφορετικές λύσεις. Αυτό θα ήταν απόλυτα καινούριο. Και ίσως η ερώτησή μου να μην είναι για σήμερα και να είναι προς την Κομισιόν, αλλά θα λάβουν υπόψη τους τα διαφορετικά στατιστικά δεδομένα. Γιατί αυτό, αυτό ήταν ο, ο συνοστισμός, αν θέλετε, το μπλοκάρισμα εδώ και χρόνια. γιατί μιλούμε για την πολιτική, το επίπεδο παρέμβασης και τα λοιπά. Είτε δηλαδή θα πάρουμε τον ΝΑΤΣ 2 και θα κοιτάξουμε τις περιοχές λειτουργίας του, ε, τις λειτουργίες πολιτικές εντός του, του ΝΑΤΣ 2 είτε θα πούμε ανεξαρτήτως σε ποιο επίπεδο ΝΑΤΣ το οποίο θα μπορούσε να είναι πολύ πιο ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, ένα σχόλιο απλώς. Μάλιστα λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσαμε να σκεπτούμε και έναν επίσημο τρόπο να συνεχιστεί πράγματι αυτή η συζήτηση γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας και τις απαντήσεις σας και θα σας περιμένουμε και στο μέλλον όταν βρούμε έναν τρόπο να διοργανώσουμε, να επισημοποιήσουμε καλύτερα τη ζήτηση αυτή και θα πάμε τώρα στο επόμενο σημείο της Μεσσίας Διατάξεως που είναι μια ανταλλαγή απόψεων ε, ε, επί γνωμοδότησης πρωτοβουλίας για την ευφυή εξειδίκευση και την μεταρρύθμιση της εδαφικής πολιτικής στην περίοδο 14-20 συμπεριλαμβανόμενου στρατηγικού προγραμματισμού για, μια, για έναν προσανατολισμό μεγαλύτερης αποδοτικότητας ε, ε, χρησιμοποιώντας τους πόρους του ECI ή στο έδαφος. Αυτά θα πρέπει να συνεισφέρουν σε μια πρώτη εξήγηση, ε, αξιολόγηση με συγχωρείτε, των μεθόδων αυτή τη στιγμή ευφυούς εξειδικεύσης και, και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα πράγματα αυτά. Ε, όπως θα θυμάστε, όπως λέγει ο παρόν κανονισμός, ε, τα επιχειρησιακά προγράμματα για την περίοδο 14-20 ε, εμπεριέχουν εξάντε προϋποθέσεις για την χρησιμοποίηση των πόρων σχετικά με τις ε, ευφυείς αυτές μεθόδους εξειδίκευσης. Ο εισηγητής μας θα μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης το Φεβρουάριο και μάλλον θα ψηφίσουμε τον Απρίλιο. Προκατακτικά βεβαίως τα λέω αυτά. Έχουμε σκιώδεις εισηγητές ε, μερικοί από τους οποίους είναι παρόντες στην αίθουσα και θα τους δώσω το λόγο για συζήτηση. Ο κύριος ε, Βαλκάρθελ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. στην συνάδελφοι. Θα γνωρίζετε ότι την προηγούμενη περίοδο εντολής με την υποστήριξη προς θεματική 1 καθορίστηκε ότι οι περιφέρειες έπρεπε να εστιαστούν περισσότερο στην έρευνα, την ανάπτυξη και στην κοινοτομία μέσω των στρατηγικών εφιούς εξειδίκευσης για την περίοδο 14-20. Οι στρατηγικές αυτές συνιστούν μια εξάντε εκ των προτέρων προϋπόθεση προκειμένου οι ευρωπαϊκές περιφέρειες να λαμβάνουν διαρθωτικά ε, πόρους των διαρθωτικών ταμείων και, των, ε, και επενδυτικούς πόρους. και αυτό πριν από την έγκριση των προγραμμάτων, το οποίο παρεμποδίζει την χορήγηση των πόρων αυτών για την επίτευξη του θεματικού στόχου, δηλαδή την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη. Και εδώ βλέπουμε τον προσανατολισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής ώστε να εστιαστεί η οικονομία αυτή ή στην καινοτομία και στην ε, Ευφύει αυτή η εξειδίκευση ώστε να γίνουν οι περιφέρειες και οι περιοχές της Ευρώπης πιο ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο πλαίσιο. Επομένως η εδαφική προσέγγιση κάθε περιφέρειας είναι κρίσιμη σημασία. Πρέπει να εστιάζεται η κάθε περιφέρεια στις δυνατότητες της ώστε να τις μεταφράζει σε μια στρατηγική αλλά με ευρύτατη γνώση του τι σημαίνει καινοτομία μακροπρόθεσμα ή μάλλον σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό ο συντονισμός μεταξύ των οντοτήτων και των φορέων πολυεπίπεδα είναι επίσης θεμελιώδους σημασία προκειμένου να επιτύχει κανείς μια αποτελεσματική υλοποίηση σε περιφερειακό επίπεδο. Από την αρχή της παρούσας περίοδου 14-20 οι ευρωπαϊκές περιφέρειες ξεκίνησαν την ανάπτυξη και την δημοσίευση των στρατηγικών του εφίους εξειδικεύσης. Τώρα, δεδομένη της σημασία του θέματος αυτού για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχω την αίσθηση ότι η εισήγηση αυτή θα μπορούσε να απαιτεί την ανάλυση της υφισταμένης κατάστασης προκειμένου να έχουμε διδάγματα για το μέλλον σε πτυχές πολύ σημαντικές όπως η ταυτοποίηση, η υλοποίηση και η αξιολόγηση των στρατηγικών αυτών. Και ο ρόλος που θα πρέπει να διαγραμματίζουν προκειμένου να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων Ευρώπη 2020. Εντός των μέσων και των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της καινοτομίας και του ρόλου που μπορούν να διαματίζουν οι στρατηγικές αυτές για την αστική, στο αστικό θεματολόγιο που θα αναπτυχθεί στου ερχόμενους μήνες υπό Ολλανδική Προεδρία και θα μετατραπεί υπό, το επερχόμενο, υπό την επερχόμενη συμφωνία του Άμστερνταμ. Αυτές είναι κάποιες από τις πτυχές που εξετάσαμε για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την ε, γνώμη αυτή και μέσω της ανταλλαγής μας απόψεων ελπίζω να έχω τις ε, απόψεις σας και τη γνώμη σας για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε καλύτερα τις ανησυχίες και τα ζητήματα που θεωρούμε υψηλής προτεραιότητας ώστε να έχουμε μια πληρέστατη γνωμοδότηση εις το τέλος. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίαση αυτή. Και τώρα, συνάδελφοι, για το λόγο. Ποιος θα ξεκινήσει. Ο κύριος Δεν είμαι σκιώδη. δεν ξέρω πού είναι σκιώδη. Α ξεκινήσουμε, δίκιο έχετε, με του σκιώδη. Ο κύριο Φαμίλτεμπουργκ, Σα ευχαριστώ. Πρόεδρα, θα μιλήσω και στη γλώσσα μου. Γιατί νομίζω ότι οι κατοχώρες αποτελούν ένα υπόδειγμα για την στρατηγική, περιφαριακή στρατηγική. Και αυτές οι στρατηγικές λοιπόν έχουν αποδείξει την αξία τους και την επιτυχία τους σε διάφορες περιφέρειες και στις κατοχώρες, στη δική μου χώρα, αλλά και εντός και εκτός της υπόλοιπη Ευρώπης. Και πάντα έχω υπόψη μου θέματα εφίους ε, καινοτομία και εξειδίκευση. σε Silicon Valley, κατεξοχήν παράδειγμα. Βασική προϋπόθεση είναι το να καταστεί προτεραιότητα η κοινοτομία για όλες τις περιφέρειες. Για παράδειγμα, για την ε, οικονομία της γνώσης, για την ανάπτυξη, για τις ε, θέσεις ε, απασχόλησης βάσει της κοινοτομίας. Πώς μπορούν αυτές να υποστηριχτούν και στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της Ευρώπης και σε διάφορες περιοχές που βρίσκονται σε φάση μεταμόρφωσης. Θα πρέπει να υπάρχει τετραπλέη ε, διάσταση, συνεργασία μεταξύ των αρχών, των ε, εργαζομένων, των εργατών, των εργαζομένων, των εργοδοτών και θα πρέπει ο στόχος να είναι να υπογραμμιστούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής. Κάθε περιοχή νομίζω ότι έχει ε, πλεονεκτήματα και μία ενδογενή αξία. Θα πρέπει λοιπόν να τα εκμεταλλεύεται. Γιατί συχνά, όταν μιλάμε για την ευφυή αυτή εξειδίκευση, γίνεται το εξή λάθος. Ε, δεν θα πρέπει να απομιμούμαστε διάφορα μοντέλα και εδώ θα ήθελα να αναφέρω και τη δική μου ε, εμπειρία στη βόρειο, στο βόρειο, στην βόρεια περιοχή του Μπράπαντα από όπου προέρχομαι και την ξέρει και την περιοχή αυτή ο κύριος Φανίστεν Ρόι ε, κοιτάμε τι γίνεται σε περιοχές υψηλής τεχνολογίας, για παράδειγμα στο Eindhoven. Και έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σε περιοχές όπου υπάρχουν πολλές εταιρείε οι οποίες πραγματικά καινοτομούν και ε, ζηλεύουμε αν θέλετε και προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε αυτά και στη δική μας την περιφέρεια. Δεν λειτουργούν όμως έτσι τα πράγματα. Πρέπει ο καθένας να κοιτάει πού έχει τη δύναμη η κάθε περιοχή. Το copyright δεν είναι right to copy, δεν είναι δικαίωμα να απομιμούμαστε. Αυτό τι σημαίνει. Όταν καταστρώνουμε στρατηγικές καινοτομίε, θα πρέπει να βρίσκουμε σε πρώτη φάση πού έγκυται αυτή η ενδογενής υπεραξία της κάθε περιφέρειας και θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι συνέργειες που μπορούν να προκύψουν μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ταμείων ε, Εθνικών Ταμείων και των Ταμείων Επενδύσεων όπως ορίζοντας, με προγράμματα όπως ορίζοντας 2020 αλλά και άλλα προγράμματα όπως το κόσμο αλλά και το Ταμείο ε, Επενδύσεων του Juncker. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και επίσης ε, κονδυλία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα ήθελα λοιπόν στην έκθεση να επικεντρωθούμε στα σημεία αυτά. Και θα ολοκληρώσω στο σημείο αυτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί τα αποτελέσματα, όπως είπε και στον αδελφός Βαλκαρσέλ, θα πρέπει να αξιολογηθούν με εντελέχεια Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τη στρατηγική ρηστρία σε όλες τις περιφέρειες και μπορεί κάποιες να μην αξιοποιούν επαρκώς και θα πρέπει να δούμε λοιπόν ε, τι γίνεται για την αξιοποίηση της γνώσης, πώς πετυχαίνουμε τη γνώση αυτή και πώς μπορούμε η γνώση αυτή μέσω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να διοχετευτεί στην αγορά και να αξιοποιηθεί μέσω υπηρεσιών και προϊόντων, μέσω κινητομιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το θέμα γιατί επενδύουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά μόνο η γνώση φυσικά ε, είναι χωρίς ε, οικονομικό αποτέλεσμα, χωρίς οικονομικό αντίκρισμα. Θα πρέπει να κοιτάμε τι γίνεται και με τα ταμεία. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ε, ποια η σχέση μεταξύ της στρατηγικής ΡΙΣ 3 και μεταξύ των περιοχών που ακολουθούν πιο τομεακή προσέγγιση και κοιτάνε πιο πολύ πώς θα ε, υποστηρίξουν τις, τους τομείς αυτούς και τις περιοχές, τις περιφέρειες οι οποίες κοιτάνε πιο πολύ τη συνολική διάσταση και θα πρέπει να κοιτάξουμε πιο πολύ και την διατομεακή συνεργασία. Και εκεί πιστεύω ότι έγινε το μεγαλύτερο δυναμικό καινοτομία. Προσβλέπω λοιπόν στη μελλοντική συνεργασία μαζί σα και με του υπόλοιπου σκιοδησίτε και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε το πώ πραγματικά οδηγεί το RIS 3 σε καινοτομία στην Ευρώπη. Αυτά, πρόεδρα και πολύ σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είστε σκιώδης οπότε σας δώσαμε περισσότερο χρόνο. Κανένα πρόβλημα. Οι άλλοι συνάδελφοι. Ο κ. Φανίστροι. Θα ehm, ook in het Nederlands eh, spreken. Ehm, de, eh, het RIS 3 heeft Θα μιλήσω στα Ολλανδικά. Σε ό,τι αφορά το RIS 3, η ιστορία είναι μακρά. Και εδώ και καιρό ε, ασχολούμαστε με τις καινοτομικές στρατηγικές της περιφέρειας. Δεν υπήρχε ερεσιμότητα αρχικά, αλλά συμπεριλαμβανόταν. όλα τα προγράμματα, όλο ο σχεδιασμό πριν από την εκτέλεση των προγραμμάτων. Και θυμάμαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα παρουσίασε τη, το 3. Ήμουν αρκετά διστακτικός, να σας πω την αλήθεια. Και έλεγα ότι μα όλοι με αυτό ασχολούμαστε. Όντως, όντως, η επικέντρωση του Ρίστρια με τις ε, δημόσιες υπηρεσίες, ε, τους δήμους, κοινότητες, τα σχολεία. Απέδωσε καρπούς. Και αυτό που επέτρεψε σε καρπούς είναι το ότι αναζητήσαμε ποια είναι η υπεραξία, ποια είναι το δυνατό σημείο της κάθε περιφέρειας. Και όχι μόνο σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ΡΙΣ αφορά την επένδυση κονδυλίων της Ένωσης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα πρέπει να ατενίσουμε και το μέλλον και να δούμε τι γίνεται με τους άλλους ε, συναδέλφους στον εκάστοτε οικονομικό κλάδο, στην αυτοκινητοβιομηχανία, σε τεχνολογίες εχμής, σε κοινωνικούς τομείς. Αυτός ο σύνδεσμος, αυτή η σύνδεση και τα έγγραφα τα οποία έλαβα και ε, τα στοιχεία με τα οποία ενημερώθηκα. Αυτές οι συμφωνίες ε, εταιρικής σχέσης. Απογοητευτήκαμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία και η τάση λοιπόν που διαμορφώνονται σε κάθε κλάδο με απασχολεί. Τι γίνεται στις ισπανικές περιφέρειες, τι γίνεται στις ολλανδικές, στις γερμανικές, στις τσεχικές, στις πολωνικές περιφέρειες. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να ερευνήσω και να κοιτάξω και τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό αφενός. Με ένα κείμενο το οποίο προσθέθηκε στον κανονισμό τότε, δηλώσαμε ότι μπορούν να αφιερωθούν κονδύλια από τη μία, να μεταφερθούν μάλλον από τη μία περιοχή, από τη μία περιφέρεια, μια αλφα περιοχή σύγκλησης, κατηγορίας 1 για παράδειγμα, σε μια άλλη περιφέρεια. Αν κάποια περιφέρεια λοιπόν διαθέτει πολλά κονδύλια, μπορεί να αποστείλει μέχρι 15% των απασχολούμενων ή των φοιτητών σε μια άλλη περιφέρεια. Μιλάμε για τεράστιο ποσό, τεράστια ποσά. Και μάλιστα με στοχοθετημένη με στοχοθετημένο προορισμό. Δεν είναι σαν το Εράσμος που πηγαίνει κανείς όπου θέλει. Όχι, πηγαίνει για παράδειγμα σε, ένα, σε μια περιφέρεια όπου υπάρχει η ίδια εξειδικευσή. Αλλά θεωρώ ότι και πάλι η φιλοδοξία είναι πολύ περιορισμένη. Δεν ε, περιοριζόμαστε μάλλον σε θέματα εφαρμογής. Θα ήθελα να γίνει ο συνδυασμός όμως αυτός ακριβώς. Όσοι εκτελούν τα προγράμματα, να τα προβάλλουν. Και ένα τρίτο σημείο το οποίο θα ήθελα να εφαρμοστεί. τα καθήκοντα του Ινστιτούτου, του Κοινού Ερευνητικού Ινστιτούτου στη Σεβελή. Για την υποστήριξη και την προώθηση του ΡΙΣΤΡΙΑ. Κυρίως στα νέα κρατή-μέλη. Πριν από κάποια χρόνια λοιπόν, με ένα πρωτικό πρόγραμμα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίξαμε και χρηματοδοτήσαμε το... την οδό προς την ε, Ευρωπαϊκή Αριστεία. Αυτά λοιπόν τα μέσα και τα κονδύλια τα δίνει το, τα αναθέτει η υπηρεσία στη Σιβήλη με αξιολογήσεις από μοτίμους, και στην προηγούμενη Ολομέλεια μάλιστα αποφασίσαμε να γίνει παράταση της χρηματοδότησης κατά δύο έτης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει και τι γίνεται. Και καλό θα είναι λοιπόν να επισκεφτούμε ως Επιτροπή το Δεκέμβριο το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο για να αισθανθούμε τον παλμό και τέλος, η ευθύης εξειδικευσή, smart specialization. Θεωρώ ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο στην αναθεώρηση της περιφερειακής πολιτικής για την περίοδο μετά το 2020. Η ευφυής εξειδίκευση περιλαμβάνει κάποια από τα στοιχεία του ορίζοντα 2020 και βλέπουμε ότι και εκεί βάσει της εξειδίκευσης της αριστείας και των εταίρων έρευνα και ανάπτυξη. Αυτό είναι ο απόκεντρος πυλώνας υποστήριξης για την τάση αυτή. Υπάρχει λοιπόν η προσέγγιση από την κορυφή προς τα κάτω από τις Βρυξέλλες και αυτή η ευφυή ε, εξειδικεύση αποτελεί μια δέσμευση από κάτω προς τα πάνω. Αν συνδυαστούν λοιπόν αυτές οι δύο μέθοδοι υποστήριξης και προγραμματισμού, αυτό ενδεχομένω να έχει μεγάλο αντίκτυπο, μεγάλη επιρροή στην περιοχή και στη φιλοσοφία, στην περίοδο και στη φιλοσοφία μετά το 2020. Μπορεί να προσθεθεί και το Stairway to Excellence Και είναι τα παλαιά κρατημέλη αυτά που κυρίως αξιοποιούν τα προγράμματα αυτά. Ορίζοντας για παράδειγμα 2020 ε, σε μεγάλο συντριπτικό ποσοστό δαπανάται στα παλαιά κρατημέλη. Θα θέλαμε λοιπόν σε ό,τι αφορά την οδό αυτή προς την αριστεία να υποστηρίξουμε νέα προγράμματα. και θεωρώ ότι αυτό θα αποτελούσε μια καλή βάση. Ευχαριστώ πολύ. Άλλοι συνάδελφοι. Κύριος Βαλκάρσελ. Συγγνώμη κύριε Βαλκάρσελ, μισό λεπτό. Έχουμε και εκπρόσωπο της Κομισιόν. Τον κύριο Μάρκ Πρεζέρ. Δεν ξέρω αν προφέρω σωστά το όνομά του. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Μια χαρά το είπατε το όνομά μου. Εκπροσωπώ την Κομισιόν. Ε, διαπραγματεύουμε το θέμα της καινοτομίας για την ευφυή εξειδίκευση τα τελευταία δύο χρόνια. Και Νομίζω ότι ε, οι, οι στρατηγικές ε, αυτές έχουν επηρεάσει την πραγματικότητα στο πεδίο πολύ. Οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες ε, είχαν, ανάγκασαν τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες να πάρουν πολύ στα σοβαρά αυτά τα πράγματα. Αλλά οι αιρεσιμότητες δεν έχουν σχέση μόνο με τη χρηματοδότηση έχουμε αρχίσει να τις βλέπουμε πια και ως ε, σχεδιασμό οικονομικής, ε, οικονομικών μεταβολών. Και κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε την ε, στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης και να πετύχουμε ρυθμού, ψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης με την καινοτομία και με προσθέμενη αξία. Βέβαια, σε ορισμένα κράτη-μέλη έχουμε έλλειψη επαρκούς διοικητικού προσωπικού, αλλά αυτή η στρατηγική δημιούργησε βελτίωση στην κατάσταση ακόμα και εκεί. Σε ορισμένε περιοχές δεν είχα περιφέρειες, δεν είχαμε ε, προσωπικό και τώρα έχουμε πολλούς ενθουσιασμένους ε, ανθρώπου που ασχολούνται με αυτά τα ζήτηματα και ακόμα και αν στην αρχή είχαμε κάποιους δισταγμούς, τώρα όλοι τα έχουν υιοθετήσει. Ε, στην αρχή νόμιζαν ότι όλα αυτά, ότι, δηλαδή ότι η ευφυή εξειδίκευση δεν ήταν τίποτα άλλο από μια γραφειοκρατική διαδικασία. Όταν όμως άρχισαν να την εφαρμόζουν, κατάλαβαν ότι είναι κάτι συγκεκριμένο, κάτι πραγματικό, κάτι που μπορεί να φέρει αλλαγή και στις επιχειρήσεις τους και στην ερευνητική τους δραστηριότητα. Οπότε επηρεάζεται όλη η κουλτούρα της έρευνας της περιφέρειας. Πρέπει να παραδεκτώ όμως ότι από τα 120 εκατομμύρια που έχουν προβλεφθεί, τα 40 είναι για την Εφή εξειδίκευση. Και οι περιφέρειες έχουν αρχίσει να βλέπουν την ανάπτυξή τους με πιο στρατηγικό τρόπο. Θέλω να πω ότι ο σχεδιασμός αφορούσε βέβαια και την προηγούμενη περίοδο, αλλά τώρα πια έχουμε μπει στη φάση της ε, εφαρμογής και των επενδυτικών σχεδίων. Έχουμε κάνει την πρώτη πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή προτάσεων και η Κομισιόν θα βοηθήσει και βοηθάει ήδη τις περιφέρειες ε, με τα κριτήρια επιλογής. Γιατί τελικά χρειαζόμαστε κριτήρια επιλογής και εκεί εμείς βοηθάμε τις περιφέρειες έτσι ώστε τα κριτήρια τους να αντικατοπτρίζουν αυτά τα οποία, τα οποία εμείς δουλεύαμε όλο αυτόν τον καιρό ε, να αναπτύξουμε. Τούτου λεχθέντος. Υπάρχει πρόοδος αλλά πολλά ακόμα θα ακολουθήσουν, ο δρόμος είναι μακρύς. Χρειαζόμαστε μια συνέχεια και συνέπεια. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι τα πράγματα δεν σταματάνε στη διαπραγμάτευση του επιχειρησιακού σχεδίου. Η συνεργατική προσέγγιση θα πρέπει να συνεχιστεί και αργότερα, θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Και αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση. Άλλη πρόκληση είναι ε, οι ιστερούσες περιφέρειες θα δουλέψουμε για αυτό το θέμα και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε τις ε, ε, χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και τις υπόλοιπε χώρες. Έχουμε δηλαδή ένα ε, χάσμα καινοτομία. Στις 18 Νοεμβρίου θα παρουσιάσουμε εδώ τα αποτελέσματα ενός μιας μελέτης που χρηματοδότησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, με την, σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μακεδονία στην Ελλάδα, 25% ε, ανεργία, διαφορετικά προβλήματα, είναι μια, πολύ, μια περιοχή με πολύ συγκεκριμένη στέρηση. ενάμιση χρόνο μετά βλέπουμε πια μια πολύ πιο δομημένη προσέγγιση. Αυτό αφορά την εφαρμογή και αυτή την προσέγγιση θέλουμε να την ε, επαναλάβουμε και σε άλλες περιοχές ε, που δυσκολεύονται να εφαρμόσουν στρατηγικές εφιούς εξειδίκευσης υψηλής ποιότητας. Τώρα, οι ε, εκ των προτέρων αιρεσιμότητες είναι λίγο διαφορετικές εδώ, διότι δεν σημαίνουν ότι χρειάζεται νομοθεσία. Όχι. Μιλάμε για μια διαδικασία αλλαγής νοοτροπίας σε ό,τι αφορά τα θέματα περιφερειακής ανάπτυξης. Γι' αυτό το λόγο ορισμένες πολλές περιοχές ε, χρησιμοποιούν τις εκ των προτέρων ρεσιμότητες για παρακολούθηση, monitoring, δηλαδή εφαρμογή της διαδικασίας ε, επιχειρησιακής, επιχειρηματικής ανακάλυψης. Ε, smart Labs, ομάδες εργασίας, focus groups, ομάδες, ε, θεματικές ομάδες, ε, εκεί η, τα πράγματα είναι πιο ευέλικτα σε ό,τι αφορά τις ε, εκ των προτέρων Η Κομισιόν θέλει όλα αυτά τα στοιχεία να λαμβάνουν την υπόψη στην εφαρμογή και, και σε ε, εργαστήρια που οργανώνουμε, workshops και σε πρακτική ε, στήριξη που παρέχουμε στο καθημερινό έργο των διαχειριστικών αρχών επιτόπου. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Κύριος ε, Βαλκάρθελ τώρα θα ήθελε να απαντήσει, να σχολιάσει. Πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σε καμία περίπτωση δεν έχω μια πρόθεση εδώ να ανοίξουμε εδώ μια συζήτηση εφόσον συμφωνούμε ότι μιλούμε για τις αναπτυγμένες περιφέρειες Ευρώπης και για τις υπόλοιπες ε, περιφέρειες που έχουν επιτύχει ένα επίπεδο, ένα ρυθμό ανάπτυξης αλλά πάντα σκεπτόμαστε την έννοια της συνοχής, της πολιτικής συνοχής και του τι σημαίνει αυτή. Όταν μιλούμε λοιπόν για μια περιφέρεια επαρκώς αν όχι υπερ-ανεπτυγμένη, πρέπει να την συνδέσουμε με συγκεκριμένες πτυχές οι οποίες επέτρεψαν αυτήν την ανάπτυξη στην περιφέρεια. Όμως εδώ μιλούμε για λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Και μιλούμε για τέτοιες περιφέρειες γιατί εξακολουθούν να υφιστάνται. Και χωρίς να εγκαταλείπουμε τους όρους καινοτομία και έρευνα οι οποίες έννοιες είναι οι πραγματικοί πυλώνες της μελλοντική οικονομικής ανάπτυξης και παρούσας μελλοντικής ε, οικονομικής ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποιες ε, υποδομές οι οποίες εμφανίζουν κενά σε αυτές τις περιφέρειες. Όμως είναι μια συζήτηση που θα μπορούσε να συνεχιστεί για το υπόλοιπο της βραδιάς και αύριο και δεν έχω τη διαπρόθεση. Τώρα, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους θερμά για τα σχόλιά τους, για τις προκαταρτικές συνεισφορές τους, γιατί μιλούμε για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, επί τη βάση της οποίας θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την, γνωμα... Ε, την... Ε, αυτή. Και θα ήθελα να, να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν και τον κύριο Βανίστελο και τους υπόλοιπους συναδέλφους, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε στο κείμενο αυτό. Ε, ο κόσμος κινείται με υπερηχητικές ταχύτητες πλέον κάθε μέρα που περνάει. Αλλά δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε, μάλλον γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε έννοιες του χθε για την ανάπτυξη του μέλλοντος. Πρέπει και οι περιφέρειες και τα κράτη-μέλη και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να παρακολουθούμε αυτήν την συνεχή ανάπτυξη και την ταχύτατη μετατροπή των συνθήκων. Ιδιαίτερα μιλώντας για καινοτομία και έρευνα, το οποίο σημαίνει συντονισμό και δεσμεύσεις σε δημόσιο επίπεδο όπως η, τράπεζα, η Τράπεζα Επενδύσεων και σε ιδιωτικό επίπεδο πάρα πολλές επιχειρήσεις που είναι έτοιμες να παρακολουθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή και να συνεισφέρουν. Τώρα, δεν έχει καθόλου άδικο ο κύριος Βανινίστελροι όταν λέει ότι οι πόροι, ο στόχος δεν είναι να δοθούν πόροι στις περιφέρειες και τίποτε άλλο. Γιατί σήμερα η αξία των οικονομικών πόρων πρέπει να επιφέρει και μια κοινωνική και εδαφική αξία και πρόοδο και να βασίζεται στις αρχές στις οποίες βασιζόμαστε όλοι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να επιτυγχάνουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και επομένως για να μην ε, μακρηγορώ, Πρόεδρε, επαναλαμβάνω ότι ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να έχουμε μια πληρέστερη δυνατή μελέτη και γνωμάτευση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει Πρόεδρος. θα περιμένουμε με ενδιαφέρον το Φεβρουάριο που θα έχουμε την πρώτη επί της ουσίας συζήτηση για την γνωμοδότησή σας. Λοιπόν, τώρα πάμε στο επόμενο σημείο της μισής διατάξεως. Έχουμε μια παρουσίαση εξωτερικής μελέτης για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία ως μέσο συνεργασίας της γενικότερης εδαφικής συνεργασίας στην Ευρώπη. Η Επιτροπή Ρέτζι ζήτησε τη μελέτη αυτή προκειμένου να εξετάσουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ιδαυγή μας συνεργασία και μετά την ε, διαδικασία ανάθεσης μέσω του Τμήματος Πολιτικής Β ανετέθη η μελέτη αυτή και εστιάζεται η μελέτη στα υφιστάμενα εμπόδια και την, ε, τις λύσεις, τις μεθόδους που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να τα παρακάμψουμε, προκειμένου έχουμε μια καλύτερη συνεργασία. Τα απορίσματα της μελέτης αυτής θα παρουσιαστούν από την κυρία Ζαμπίνε Τσίλμα, την δόκτωρα Ζαμπίνε Τσίλμα μάλλον, η οποία είναι επικεφαλής σύμβουλος και έχουμε επίσης εδώ εκπροσώπους της Επιτροπής των Περιφερειών και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Κοτέρ της Επιτροπής των Περιφερειών. Έχουμε τον κύριο Κατάνιο και έχουμε και τον πολιτικό συντονιστή της πλαθών CGTC της Επιτροπής των Περιφερειών που είχε ηγηθεί σεμιναρίου εργαστηρίου επί του θέματος αυτό σήμερα. της ευρωπαϊκής ε, λοιπόν αυτής ε, του ευρωπαϊκού φορέα της εδαφικής συνεργασίας. Παρακαλώ. Αγαπητέ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, εισαγωγή και για την πρόσκληση να σας παρουσιάσουμε αυτή τη μελέτη. Θέλουμε να προωθήσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρώπη και θα σας παρουσιάσω λοιπόν τους στόχους της μελέτης καταρχάς, ε, αναφέρατε κάποιους εξ αυτών και θα σας αναφέρω και τα σχετικά εργαλεία προτού επικεντρωθούμε στα απορίσματα της ε, έκθεσης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το δυναμικό συμβολής στην ε, πολιτική συνοχή. Σε ό,τι αφορά και την εξωτερική ε, πολιτική. Προσπαθήσαμε λοιπόν και μας δίθηκε να εκτιμήσουμε το ρόλο του EGTC στην πολιτική συνοχή και στο ETC. Αυτός ήταν ο αρχικός στόχος και ο δεύτερος στόχος ήταν η ανάλυση των ρόλων που ενδεχομένω έχουν τα ETC στην πολιτική γειτονία και ιδιαίτερω για τι αποκεντρωμένε περιοχές. Το εργαλείο αυτό του EGTC δημιουργήθηκε το 2006 με τη σχετική νομοθεσία και ως σκοπό είχε να ενισχύσει την περιφερειακή συνεργασία. Αυτός ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας αποτελεί λοιπόν ένα εργαλείο, ένα νομικό εργαλείο εντός της πολιτικής συνοχής και πέρα από την πολιτική συνοχής. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δράσει υπό μία ενότητα και υπό ένα όνομος όμιλος. Είναι μεγάλη έως τώρα η ποικιλία των διαφόρων οργανισμών που εντάσσονται στον όμιλό μας. Αλλά σπάνια χρησιμοποιούνται για τον αρχικό τους στόχο. Με την τροποποίηση του κανονισμού το 2013 διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφική Συνεργασία και ενισχύθηκε η πτυχή της σύνοχή, αναφέροντα συγκεκριμένα το σεβασμό των κανονισμών και των διαφόρων κανόνων που μπορεί να ισχύουν και των διαφορετικών ρόλων που μπορεί να έχει ο Ευρωπαϊκό Όμιλο Συνταφική Συνεργασία στην πολιτική συνοχή. Παρόμοιοι είναι οι στόχοι και τα καθήκοντα του ομίλου. Έχουμε διαφορετικά θέματα, αλλά και κάτι άλλο που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στις συστατικές συνθήκες το, ο βαθμός λεπτομέρειες για την επιτεύξη στόχων είναι σε μεγάλο βαθμό διαφορετικό. Παρά την τροποποίηση λοιπόν του κανονισμού εξακολουθούν να υφίστανται πολλές προκλήσεις για την περίοδο ιδρύση ενό Ευρωπαϊκού Ομίλου Δακτική Συνεργασίας. Και επίσης ε, Διάφορες ε, αλλαγές προκύπτουν και διαφορές προκύπτουν κατά τη λειτουργία του EGTC. Λόγω της εφαρμογής, λόγω της λειτουργίας, ε, αλλά λόγω και αβεβαιοτήτων, έλλειψης ε, γνώσεων κτλ. Και από πολλά, και αυτό ξέρετε από πολλούς παράγοντες με τους οποίους έρχονται αντιμέτωποι τα EGTC. Κατά το παρελθόν τα EGTC δεν έχουν αξιοποιήσει τους πόρους για να εκτελέσουν ε, τέτοια προγράμματα και αυτό για διάφορους λόγους, αλλά πρόσφατα έχει αυξηθεί η αξιοποίησή τους. Έχουμε λοιπόν διάφορα τέτοια προγράμματα ETC ε και κάποια EGTC ε συμμετείχαν και στην κατάρτιση των λειτουργικών προγραμμάτων. Η πολιτική συνοχής και η σχετική στόχη στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με τα θέματα τους τομείς εφαρμογής που καλύπτουν οι EGTC και επί της αρχής για όλους τους στόχους της πολιτικής συνοχής υπάρχουν και ανάλογα EGTC τα οποία ασχολούνται σε διαφορετικούς βαθμούς με τους στόχους αυτούς και εδώ βλέπουμε κάποια κάποιες θεματικούς στόχους για το περιβάλλον, τις μεταφορές, την παιδεία και το καθεξής. Και ως εκ τούτου τα EGTC τα οποία εξετάσαμε σε βάθος δηλώνουν ότι θέλουν και στο μέλλον να συνδράμουν σε διάφορους θεματικούς τομείς ακολουθώντας ενοποιημένες προσεγγίσεις σε τέτοια θέματα. Επίσης, θέλουν να αξιοποιήσουν καλύτερα τα κονδύλια και την απορρόφηση των κονδυλίων για να εκπληρώσουν τα προγράμματα και να μπορούν να αξιοποιήσουν όλες τις ε, δυνατότητες. Παρά όλες αυτές τις ε, εξελίξεις δεν αναφέρονται ιδιαίτερα στα λειτουργικά προγράμματα τα HDC. Και μάλιστα σπάνια αναφέρονται τέτοια HDC. Μόνο συγκεκριμένα αν αναφέρονται στην ε, προγραμματική περίοδο και αναφέρονται σε κάποιες περιπτώσεις τα λειτουργικά προγράμματα τα EGTC και τα ETC τα οποία χρησιμοποιήθηκαν. Μόνο στο λειτουργικό πρόγραμμα του Λουξεμβούργου εμείς εντοπίσαμε τέτοια, τέτοιες εξαιρέσεις. Σε ό,τι αφορά την εξωτερική συνεργασία, εδώ θα βρείτε συνοπτικά όχι μόνο τη συνεργασία με τις γειτονικέ χώρες και τις χώρες προσχώρησης, αλλά και τις αποκεντρωμένες περιφέρειες. Δεν διαπιστώνουμε να υπάρχουν EGTC με μέλη από τέτοιες χώρες ή από εξόχως αποκεντρωμένες περιφέρειες. Σε ό,τι αφορά τις γειτονικέ χώρες, ε, Γίνονται πολλές συζητήσεις, αλλά ως τώρα καμία δεν έχει πραγματοποιηθεί για διάφορους λόγους, κυρίως γεωπολιτικές αβεβαιότητες, οι οποίες προέκυψαν ε, προβλήματα με τις κυβερνήσεις. Οι πιο πολλά υποσχόμενες προπτικές είναι από την Ελβετία, όπου έχουν δρομολογηθεί διάφορες ε, εξελίξεις, αλλά δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί και στην περίπτωση αυτή. Και για θέματα περίπλοκης ε, της εφαρμογής σε ό,τι αφορά τις εξόχως περιοχές ως τώρα υπάρχει μια προσέγγιση η οποία έχει δρομολογηθεί στο ενίσο του Σαν Μαρτάν και κοιτώντας τα συνολικά ευρήματα και πορίσματα για τη συνεργασία. Έχουμε την εντύπωση ότι οι δυνατότητες και οι συνέπειες της χρήσης των EGTC δεν είναι ευρέως γνωστές ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε και στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και συχνά δε φαίνεται ότι υπάρχει και έλλειψη θεσμικών ικανοτήτων προκειμένου να ξεπεριστούν τα σχετικά εμπόρια. Όπως σας είπα έγινε η ανάλυση φέτος την Άνοιξη και έως τότε ήταν πολύ περιορισμένη εμπειρία, η εμπειρία μας με την τροποποιημένη νομοθεσία. Άρα δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε πραγματικά και ουσιαστικά τα αποτελέσματα της αναθεώρησης της, νομολογίας, της νομοθεσίας. Ωστόσο, από την παρούσα προοπτική εξακολουθούν να υφίστανται οι δυσκολίες αν και αυτές ενδεχομένω να ξεπερνάν τον κανονισμό του EGTC και να οφείλονται σε διαφορετικούς λόγους. Και επειδή δεν είναι καθοριστική η αξιολόγηση της ε, νομοθεσίας EGTC, είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο η εφαρμογή στην εκατότητα χώρα για την εφαρμογή και τη λειτουργία των EGTC παρά την αναθεώρηση της νομοθεσίας δεν έχει επηρεαστεί ουσιαστικά η αντιμετώπιση από τις εθνικές αρχές. Έλλειψη γνώσεων, επιφυλακτικότητα διαπιστώνουμε σε πολλές χώρες και περιφέρειες. Τέλος, ο τροποποιημένος κανονισμός EGTC επισημαίνει ότι το να αξιοποιηθούν τα EGTC για την παροχή υπηρεσιών οικονομικού ενδιαφέροντος προαπαιτεί το να λάβουμε υπόψη και να συνειδητοποιήσουμε το δυναμικό που περιέχεται στον κανονισμό για τα EGTC και προφανώς αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το πετύχει μόνο ο κανονισμός για το EGTC και ίσως εδώ η Λουξιμοργιανή Προεδρία να μπορέσει να μας ανοίξει ναι, οδούς. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω με τον τρόπο αυτό να σας παρουσίασα έστω και συνοπτικά αυτή την έκθεση που νομίζω ότι φτάνει τις 80 σελίδε αν δεν κάνω λάθος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για αυτήν πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Περνάμε σε ανταλλαγή απόψεων, ερωτήσει. Μας απομένουν 25 λεπτά. Παρακαλώ, έχει λοιπόν πάνω από πέντε λεπτά να παρέμβαση. Ποιος θέλει να ξεκινήσει, ο κύριος Τσέλερ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Καταρχήν να, να χαιρετήσω τον κύριο Κατάνιο. Έχουμε εργαστεί για, μαζί με την Επιτροπή των Περιφερειών για ένα συνέδριο διήμερο για την διασυνοριακή συνεργασία. Και είχαμε μιλήσει ιδίως για την εφαρμογή αυτού του νέου εργαλείου που έχουμε του Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας και το οποίο μας απασχολεί σήμερα. Το ανέφερα λοιπόν διάφοροι συνάδελφοι και το γεγονό ότι έχουμε μαζί μας σήμερα ε, τόσο λίγου συναδέλφου, ελπίζω να μην σημαίνει ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ομιλητευτική Συνεργασία θα λάβουν τόσο περιορισμένη προσοχή όπω και από τι κυβερνήσει μα, γιατί εξακολουθεί να, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια. Συχνά, ξέρετε, αυτό το GTC αποτελεί ε, ένα αρκετά δυσάρεστο αντικείμενο για τις κυβερνήσεις και για τις αρχές και όπως επιβεβαιώνεται και από την Επιτροπή Ρέτζη, είναι ένα άγνωστο, ένας άγνωστος τομέας. Και θα ήθελα να σας παρουσιάσω ποια είναι το ιστορικό. Ποιος ήταν, ποια ήταν η αφορμή για τους ευρωπαϊκούς ομίλους με την εδαφική συνεργασία. Προήλθε αυτό από την Επιτροπή των Περιφερειών και η περιφέρειες ως νομικές εντότητες ε, περιμένουν να έχουν μια τέτοια ευκαιρία για την διασυνοριακή συνεργασία. Γι' αυτό λοιπόν ζήτησα να, να διευκολυνθεί το έργο τους ε, της ε, διασυνοριακής συνεργασίας και αυτό γιατί μιλάμε μεν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλές περιπτώσεις για ίσους όρους ανταγωνισμού, αλλά σε διάφορες περιπτώσεις υπάρχουν εθνικά δίκαια 28 κρατών μελών και μάλιστα αυτά τα δίκαια συχνά διαφέρουν και σταματούν στα σύνορα της κάθε χώρας ασφαλώς. Και αυτό δυσχεραίνει, μη σας πω κάνει και αδύνατη συνεργασία σε κάποιες περιπτώσεις. Και από εκεί λοιπόν προέκυψε η ιδέα του να δημιουργηθεί ένα νομικό εργαλείο το οποίο θα επιτρέπει τη συνεργασία θα οργανώνει τη συνεργασία και η τότε επίτροπος Ντανούτα Χούμπνερ ήταν εκείνη η οποία πρότεινε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Κοινοβούλιο την πρόταση αυτή και το τελευταία θητεία, ε, στην τελευταία θητεία αποφασίσαμε και κρίναμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι διαβριμενο κανονισμό με διαβριμένες δυνατότητες σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής διευρύνθηκε, αλλά προβλέφθηκαν και δυνατότητες συνεργασίας και περιλαμβάνουν πλέον και δημόσιες κοινοφελείς υπηρεσίες, δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιες εταιρείες, ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες μπορούν να συμμετέχουν πλέον για την εφαρμογή των εργασιών αυτών και να μην ε, χρησιμοποιείται επίσης αυτό το εργαλείο μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διασυνοριακή συνεργασία, αλλά και σε συνεργασία με τα γειτονικά κράτη της Ένωσης, όπως αναφέρθηκε. Ναι, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα και θα πρέπει να τονίσω, επειδή συμμετείχα και στους τριμερεί διαλόγου, ότι η αντίσταση ήταν μεγάλη από πλευρά των κρατών μέλων λες και με ζήλια παρακολουθούσαν τα κρατημέλη να μην δώσουν υπερβολικά μεγάλες αρμοδιότητες και ελευθερίες στις ε, περιοχές κοντά στα σύνορα. Γιατί φαίνεται ότι αυτό επικρατεί ως ντροπία στις πρωτεύουσες. Κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά τους ε, φορείς ε, επιτόπου οι οποίοι είναι συνηθισμένοι στη συνοριακή συνεργασία, τα προγράμματα ίντερνετ και το καθεξής. Μεταξύ αυτών δεν υπάρχει επαρκής σαφήνεια για το ότι είναι νομικό εργαλείο, το οποίο δεν υποχρεώται φυσικά κανείς να αξιοποιήσει και να χρησιμοποιήσει, αλλά μπορεί αν θέλει. Έτσι λοιπόν μπορούν να δημιουργηθούν α, ε, θεσμικοί φορείς, να προσλάβουμε προσωπικό, να αξιοποιηθούν τέτοιες δυνατότητες που θα διευκολύνουν την εργασία, ιδιαίτερα στις διασυνοριακές περιοχές. Κάποιοι τα καταφέρνουν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις νομίζω ότι υπάρχουν ελλείμματα και στην ενημέρωση και στην επικοινωνία. Η έκθεση, η μελέτη την οποία έχουμε στη διάθεσή μας, νομίζω ότι υποδεικνύει ακριβώς τα αδύναμα σημεία τα οποία θέλαμε να απαλείψουμε στον τελευταίο τριμερή διάλογο και όπου αποτύχαμε. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε την εμπειρία που έχουμε σήμερα θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις τελευταίες εμπειρίες προκειμένου αυτά να μπορέσουν να μπουν και στην ενδιάμεση θεώρηση στη συζήτηση και να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε τη διαμόρφωση αυτού του νομικού εργαλείου. Ιδιαίτερα σε μια χρονική στιγμή όπου βάσει λόγω και των πρόσφατων περιστατικών ε, πάλι ψώνονται φράχτες, πάλι ε, μιλάμε για ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν καθημερινά τα κρατημέλη. Ή συνεργασία μεταξύ των ε, περιφερειών αυτών, των διασυνοριακών αυτών περιφερειών, δεν πρέπει να επιβαρυνθεί λόγω των ε, συνθήκων. Πρόκειται για ένα καλό εργαλείο, αλλά διαπιστώνω ότι αυτές οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης δεν αναφέρουν καν τα EGTC. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι είναι δικαίωμα του καθενός να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία, μιας και περιλαμβάνονται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά παρόλα αυτά διαπιστώνουμε ότι δεν αναφέρονται σε πολλές περιπτώσεις καν στα λειτουργικά προγράμματα τα EGTC. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την μελέτη και για την απόπειρα να δώσουμε σάρκα και οστά σε αυτό το νομικό εργαλείο και να χρησιμοποιηθεί επαρκώς αυτή η πλατφόρμα Και σε κάθε περίπτωση από πλευρά τη Επιτροπή μα θα πρέπει να συνεχίσουμε προ την κατεύθυνση αυτή για την ενίσχυση περαιτέρω τη διασυνοριακή συνεργασία και για την κατάργηση και την απαλήφη των γραφειοκρατικών εμποδίων, καθώ και την επίλυση των σχετικών παρανόησεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριο Σόλμπριχτ. Ίσως θα ήταν κρίσιμο να δούμε λίγο ε, ορισμένα στοιχεία. Ήμουν ο πρώτος εισηγητής για τους ομίλους εδαφικής συνεργασίας, οπότε να κάνω μια ε, ιστορική αναδρομή. Ε, η ιδέα προήλθε κατά 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καμία σχέση δεν είχαν οι τοπικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκείνη την εποχή ε, ήθελε να διαθέτει ένα ευρωπαϊκό όργανο, ε, εργαλείο που το, ονομούσαν, το, το ονομάζανε GCC στην αρχή. Ο Ζων Σαρλέγκ μας εξηγούσε ε, ότι είναι κάτι πολύ απλό, πολύ ευρωπαϊκό και θα το δεχτούν όλοι πολύ εύκολα. Εγώ είχα επιφυλάξεις, αλλά μου έλεγε ότι προέρχομαι από καινούριο κράτος μέλους και δεν καταλαβαίνω την Ευρώπη. Και ότι θα το δεχόντουσαν πολύ εύκολα. Εγώ εξ αρχής είπα, έλεγα, πρόκειται για συνταγματικό θέμα, δεν είναι τυπικό. Έχει νομικές συνέπειες αυτό το εργαλείο, γιατί τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη με δύο διαφορετικούς κανονισμούς της αγοράς εργασίας, δύο διαφορετικούς οικονομικούς κανονισμούς κλπ. δημιουργούσαν ε, επιπλοκές. Γι' αυτό το λόγο το αλλάξαμε και το απλοποιήσαμε. Για να το απλοποιήσουμε τι κάναμε. Καταφέρουμε να εξηγήσουμε στην Κομισιόν, να την πείσουμε ε, από EGCC να γίνει EGT δηλαδή εδαφική συνεργασία και όχι διασυνοριακή συνεργασία όπως ήταν στην αρχή, όχι cross-border αλλά territorial cooperation. Η Επιτροπή των Περιφερειών από την αρχή διαφωνούσε. Γιατί? Γιατί φόντουσαν ότι το καινούριο αυτό εργαλείο, το καινούριο μέσο θα τους αφαιρέσει την ε, διασυνοριακή συνεργασία που λειτουργούσε πολύ καλά. Τις ε, ευρωπεριφέρειες κλπ. κλπ. Φοβόντουσαν ότι αυτά τα, αυτό το μέσο θα αναλάμβανε, θα, μάλλον θα έπαιρνε αυτή την αρμοδιότητα από την Επιτροπή των Περιφερειών και θα την ανέθετε σε κάποιον άλλο φορέα. Υπουργεία ή οτιδήποτε άλλο. Εμεί του εξηγήσαμε λέγοντα ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το καινούργιο μέσο για την υφιστάμενη συνεργασία. Δεν ήταν και πολύ σίγουροι ότι θα λειτουργήσει έτσι, αλλά του προτείναμε να αναλάβουν η Επιτροπή των Περιφερειών την παρακολούθηση του καινούριου μέσου. Δέχτηκαν και άρχισαν να κάνουν το, την παρακολούθηση. Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλά τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί ακόμα. Γιατί η νομοθεσία είναι περίπλοκη, οι συμφωνίες είναι περίπλοκες, οι διοικητικές ικανότητες ήταν διαφορετικές. Το πιο δύσκολο πράγμα εκείνη τη στιγμή ήταν ότι το Συμβούλιο, το Συμβούλιο συμφώνησε με το μέσο αυτό υπό έναν όρο ότι δεν θα δημιουργηθεί χωρίς τη Συμφωνία των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων. Γιατί η αρχική ιδέα ήταν οι τοπικές αρχές να δημιουργούν ομίλους εδαφικής συνασίας και να ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω δημοσίευσης στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία τέτοιων ομίλων. Όμως ε, τότε είχαν στο μυαλό τους το, τα προβλήματα μεταξύ Σλοβακίας και Ουγγαρίας και άλλων περιοχών όπου πολιτικά θα ήταν εκρηκτικό οι τοπικές αρχές να δημιουργούν τέτοιου ομιλού ομίλους ε, ε, χωρίς γνώση των κυβερνήσεών τους. Οπότε αυτό ήταν ο όρος που βάλε το Συμβούλιο οι όμιλοι εδαφικής να δημιουργούνται κατόπιν συμφωνίες των κυβερνήσεων. Οπότε εκεί Έχουμε διαδικασίες πολύ πιο περίπλοκες και χρειαζόμαστε και κατάλληλες διοικητικές ικανότητες. Υπάρχει όμως συνεργασία, διασυνορική συνεργασία και γι' αυτό το λόγο ήταν σημαντικό αυτή η συνεργασία που ήδη υπάρχει να γίνει εδαφική συνεργασία. Να κάνουμε δηλαδή ένα νομικό πείραμα. Για παράδειγμα τους, τους είπα ε, συνεργασία για την κατασκευή της γέφυρας και αυτοί ξέρανε γέφυρα, ποια γέφυρα μιλώ, ε, για ποια γέφυρα μιλούσα ή ε, για συνεργασία για την κατασκευή ενός νοσοκομείου στα σύνορα. Ε, δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσει η αντίδραση γιατί οτιδήποτε δεν είναι εθνικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπλοκο. Οτιδήποτε διασυνοριακό είναι δύσκολο. Ε, προσπαθήσαμε να το σπρώξουμε λοιπόν για να λειτουργήσει αλλά ορισμένες ανησυχίες, μάλλον βλέπουμε σήμερα την ε, συνέπεια ορισμένων ανησυχιών που είχαν εκφραστεί από παλιά, την αρχή. Είναι σημαντικά όλα αυτά που λέω γιατί είναι ιστορική μνήμη. Έτσι καταλαβαίνουμε τη σημερινή κατάσταση. Στην πρώτη συνάντηση του Συμβουλίου, να σας θυμίσω, τα δύο τρίτα των κρατών μελών διαφωνούσαν και έτσι είχα πει εγώ στην Κομισιόν, έτσι λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, βλέπετε πόσο εύκολα, <laughs> βλέπετε πόσο εύκολα ε, απορρίφθηκε, ενώ εσείς νομίζατε ότι θα εγκριθεί πολύ εύκολα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τσέλα για κάποια σχόλια για να συνεχίσουμε μετά. Πολύ καλά τα περιέγραψε ο Γιάννη. Και επαναλαμβάνω. ανεξάρτητα από το που προέρχεται η αντίσταση. Το θέμα είναι κατά πόσο θα αποδεχτούμε την κατάσταση αυτή όσο έχει. Ναι, μεν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια πρόταση για την δεσμευτική συνεργασία, αλλά επαναλαμβάνω, ξέρω ότι ανάγκη για ένα τέτοιο εργαλείο προέκυψε από τι ίδιε τι περιφερειέ, από κάποιες έστω, οι οποίες εξέφρασαν αυτή την επιθυμία στα πλαίσια της Επιτροπής των Περιφερειών και γι' αυτό λοιπόν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία στην Επιτροπή των Περιφέρειων. Τα μεγαλύτερα προβλήματα όμως δυστυχώ, σε αυτή τη φάση τα έχουμε στα συνορα γερμανια Γερμανίας-Πολωνίας. Είναι πραγματικά εξωφρενική η κατάσταση. Αφενός έχουμε ε, τοπικού άρχοντε οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να ε, αφήσουν κατά μέρο κάποιες αρμοδιότητες σε άλλους, το οποίο δεν ισχύει και αφετέρου τη δυνατότητα συνεργασίας με τους συναδέλφους ε, από την άλλη πλευρά του, του, των συνόρων. Είτε πρόκειται για α, προγράμματα συγκοινωνία, δημοσίων υπηρεσιών, ε, εκπαίδευση, ό,τι και να είναι, πάντα υπάρχει ο φόβος ότι κάτι θα χάσουν. Και παράλληλα, όπως είπε ο Γιάνν, τα προγράμματα αυτά και η μορφή συνεργασίας πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά στις πρωτεύουσε και μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα τέτοια οργάνωση. Στην Πολωνία υπεύθυνη είναι η εθνική κυβέρνηση, η κεντρική κυβέρνηση. Στην Γερμανία είναι η κυβέρνηση των κρατήδιων, άρα δεν υπάρχει αντιστοιχεία μεταξύ των επιπέδων, γιατί ε, το Πολωνικό λέει, Υπουργείο δηλώνει ότι θα μιλήσουμε μόνο με την Εθνικό της Υπουργεία της Γερμανίας και τελικά υποφέρουν και πλήττονται τα προγράμματα τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Και μιλάμε για απλά πράγματα. Έχουμε διάφορες πόλεις, για παράδειγμα, οι οποίες ε, ε, ουσιαστικά χωρίζονται από τα εθνικά σύνορα. Φραγκφούρτη, Όντρες Τσούμπιτσε, για παράδειγμα, επειδή έχουν ένα πανεπιστήμιο που είναι και στην πολωνική πλευρά αλλά και στη γερμανική πλευρά, και ήθελα να έχουν λοιπόν μια σύνδεση με το ηλεκτρικό ή με το λεωφορείο για να μπορούν οι φοιτητέ να πηγαίνουν από τη μία πλευρά στην άλλη. Και γι' αυτό λοιπόν θέλανε έγκριση και από το ΠΟΤΣΤΑΠ και στην Πολωνία θέλανε και χρειαζόντουσαν την έγκριση από το Πολωνικό Υπουργείο. Πέντε χρόνια πήρε μέχρι ότου εγκριθεί αυτή η γραμμή του λεωφορείου, η οποία σήμερα χρησιμοποιείται πιο πολύ από κάθε άλλη. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι χρειάζεται κατεπηγόντως να αναλάβουμε δράση προκειμένου να ξεπερνούνται τέτοια προβλήματα σε περιοχές κοντά στα σύνορα. Και πλέον οι Ευρωπαϊκή Όμιλη Εδαφική Συνεργασία δεν απειλούν σε τίποτα τι ήδη υφιστάμενε μορφέ συνεργασία. Αντιθέτω, αποτελούν ένα νομικό εργαλείο, δεν είναι εργαλείο υποστήριξη. Με το εργαλείο λοιπόν αυτό είναι δυνατόν με ευρωπαϊκό δίκαιο να διευκολυνθεί η συνεργασία όπου δεν το επιτρέπει αυτό ενδεχομένω η εθνική νομοθεσία προκειμένου και να σημειωθεί η πρόοδο. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Ο, κ... ο κ. Βαλνίστερο έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Κοιτώντα την ε, έκθεση αυτή και την ε, σχετική παρουσίαση και επεξήγηση, το θέμα είναι κατά πόσον μα ικανοποιεί η εξέλιξη και η ανάπτυξη του μωρού. Α το αναφέρουμε έτσι. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε ότι αναπτύσσεται σωστά. Αλλά πέρα από το εργαλείο αυτό υπάρχει πολύ πιο πολλή συνεργασία από την μία περιοχή στην άλλη. Έχουμε πάρα πολλά καλά παραδείγματα τέτοια διασυνοριακή συνεργασία. Τη στιγμή τη ε, των ε, νέων κρατών μελών. Υπήρχε ανάγκη μεγαλύτερης και πιο γρήγορης συνεργασίας. Και αυτό γίνεται με νομικά μέσα. Αν υπάρχουν νομικά μέσα, δεν χρειάζεται 20 χρόνια. Μπορεί κανείς ε, να κλείσει συμφωνίες με τα διάφορα κράτη-μέλη πολύ πιο γρήγορα, να ορίσει αρμοδιότητες σε κάθε περιφέρεια. Και ίσως και να υπερτιμήσαμε τις ικανότητες μας για τις δυνατότητες που είχαμε. Κοιτάξτε, εγώ τότε ήμουν στη συνέλευση των Ευρωπαϊκών Συνοριακών Υπηρεσιών και κάναμε και σχετική γνωμοδότηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά που διαπιστώνουμε τώρα είναι καλά παραδείγματα. Αυτός ο ενθουσιασμός της πρώτης περίοδου υπάρχει ακόμα. Για παράδειγμα μεταξύ Βελγίου και Ολλανδίας, όπου υπήρχε ήδη μια συμφωνία για τα έργα που χρειάζονταν να γίνουν. Δίνεται λοιπόν μια επιπλέον διάσταση στην εργασία από τον τρόπο αυτό. Όταν εντός του κράτους μέλους δεν επικρατεί θετική διάθεση, είναι σχεδόν αδύνατο να το πετύχουμε. Στην Ολλανδία, η συνεργασία μεταξύ Ολλανδίας και Βελγίου, στην περιοχή Λίμπουργκ και μεταξύ της Γερμανίας, υπάρχουν και έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχα εργαλεία και μέσα από τα κρατήδια, από τη Βαλονία. Έχουν προκύψει λοιπόν τέτοια εργαλεία, αλλά δεν ονομάζονται ομίλος οδαφικής συνεργασίας. Δεν θέλουν να τα πούνε έτσι απλά. Δεν θέλουν να τα πούν ή. GDC. Και παρουσιάστηκαν ως κάτι το οποίο ανέπτυξαν τα κράτη-μέλη από μόνα τους. Δεν το λέμε έτσι, το λέμε αλλιώ. Το ίδιο πράγμα όμω είναι. Γι' αυτό λοιπόν και στην παρουσίαση σα είπατε ότι δεν αναφέρονται στα λειτουργικά προγράμματα καν η Ευρωπαϊκή Όμιλη Εδαφική Συνεργασία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο σίγουρα μας χρησιμεύει. Είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρήσουμε ότι με τον τρόπο αυτό και με τη χρήση του εργαλείου αυτού θα μειωθεί η εδαφική και διασυνοριακή συνεργασία. Όχι. Πάρα πολλά συμβαίνουν και γίνονται διασυνοριακά. Και κοιτώντα και τις εξελίξεις και την ανάπτυξη της συνοχής, την περιφερειακή συνεργασία και την περιφερειακή συνοχή, ένα από τα στοιχεία είναι ότι αυτή η διασυνοριακή πτυχή εξακολουθεί να έχει ύψη σημασία. η συνεργασία θα παραμείνει ύψης της προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν προσπαθήσουμε να προβλέψουμε τι θα γίνει τα επόμενα 20 χρόνια, σίγουρα θα παραμείνει αυτό ένα πολύ σημαντικό κατεξοχήν ευρωπαϊκό εργαλείο. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Κατάνιο συντονιστής του EGTC της σχετικής πλατφόρμας από πλευρά της ε, Επιτροπής των Περιφερειών. Ίσως θα θέλετε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για το σημερινό σεμινάριο για την πρωτοβουλία EGTC. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία της ε, διερμηνίας για να μιλήσω στα Ιταλικά. έχοντας ακούσει με ενδιαφέρον την ε, εξιστόρηση αφήγηση του Γιάνν Όλμπριχτ που θεωρώ ότι περιέγραψε πολύ σωστά κάποια από τα βασικά προβλήματα και τις πολιτικές στοιχές που διέπουν το θέμα αυτό. Εγώ θεωρώ ότι πίσω από τον όμιλο αυτό που είναι το μοναδικό νομικό πλαίσιο που έχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι κοινοτικοί φορείς για να αναπτύξουν τη διασυνορική συνεργασία. Υπάρχει η αντιπαράθεση μεταξύ δύο διαφορετικών οραμάτων για την Ευρώπη. Μία top-down και εδώ εξηγούμε ότι εδώ πρόκειται για μια πρωτοβουλία της ε, Κομισιόν στην οποία ανέφεραν αντίθεση οι τοπικοί φορείς όπως λέει ο, ο κ. Όλμπριχτ και μια άλλη εντο αλλου άλλου οράματος bottom-up. <clears throat> Αν θέλουμε δηλαδή να στηριχθούμε στις πρωτοβουλίε και στι δραστηριότητε των τοπικών και περιφερειακών φορέων θα χρειαζόμασταν πολύ περισσότερες δομέ αντίστοιχε. με το EGTC. Είχαμε και ένα εργαστήριο και τη συμμετοχή του ομίλου στην ε, ευρωπαϊκή συνεργασία και στη διασυνεργειακή συνεργασία που, το οποίο έφερε στο φως και πολλές από τις τεχνικές δυσκολίες και άλλες δυσκολίες. Όμως πίσω από όλα αυτά υπάρχει, επαναλαμβάνω, ένα πολύ σημαντικό πολιτικό θέμα. Η Επιτροπή των Περιφερειών επενδύει στη θεματική αυτή θεωρώντας το EGTC ένα στρατηγική σημασίας μέσων ώστε να έχουμε μια πραγματική συμμετοχή τοπική στη διασυνοριακή συνεργασία και στην ανάπτυξη. Και για τον λόγο αυτό έχουμε αναπτύξει μια πλατφόρμα υπό το EGTC που τώρα έχω την ευθύνη της μάλιστα, της διαχείρισής της που παρακολουθεί την υλοποίηση της εθνικής νομοθεσίας προσπαθεί να αναπτύξει την επιφάνεια του μέσου του ομίλου και να ταυτοποιήσει και κάποια προβλήματα, κάποια σημεία συμφόρησης και προσπαθούμε να διατηρήσουμε και ένα αρχείο αν θέλετε όλων των ομίλων τοπικών φορέων όπου αντίστοιχα ενημερώνουν την Επιτροπή των Περιφερειών και καταχωρίζονται αν θέλετε επισήμως. Έχουμε λοιπόν 56 συνολικά ομίλους στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, η GTC, από, που εκπροσωπούν 500 φορείς από 26 χώρες. Είναι σημαντικός ο αριθμός, αλλά δεν είναι εντυπωσιακός. Και αυτό ίσως θα μπορούσε να μας δημιουργήσει κάποιες σκέψεις για τους περιορισμούς και τις δυσκολίες. Και τον περασμένο Σεπτέμβριο η Προεδρία του Λουξεμβούργου ξεκίνησε μια πρωτοβουλία επανεξέτασης και των νομικών μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να υποστηριχθεί η διασυνοριακή συνεργασία και τον Οκτώβριο ενέκρινε και μια γνωμοδότηση ε, όπου αναπτύσσεται η αναγκαιότητα μιας επικαιροποίησης νομοθετικού πλαισίου. Τώρα και για λόγους ε, χρονικού περιορισμού, ε, εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω τις δυσκολίες που εμείς καταφέραμε να εντοπίσουμε. Καταρχάς οι τροποποίησεις που έχουν επέλθει στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο των GTC που απλούστευσε τις διαδικασίες που ήταν το αποτέλεσμα μια καρποφόρα ε, συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τσέλα που ήδη από τότε ήταν εισηγητή μαζί με την κυρία Ντανούτα Χύμνα και με την πρόεδρο Μιχαήλοβα είχαμε ξεκινήσει μια εξίσου θετική και ίσως ακόμα περισσότερη συνεργασία. Εν πάση περιπτώσει κάποιες χώρες όμως δεν συμφωνούν προς τις τροποποίησει αυτέ και έτσι αυτό που κάνουν είναι ότι απλά δεν τις υλοποιούν. ούτε το ίμιση των εθνικών αρχών δεν έχει προχωρήσει στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για του CGTC και θα έπρεπε να το έχει κάνει μέχρι τον Ιούνιο πέρυσι. Υπάρχει επίσης μια έλλειψη συμμετοχής των υφισταμένων EGTC στην προετοιμασία των ε, επιχειρησιακών προγραμμάτων. Άρα αυτό είναι ένα... Το πλαίσιο δηλαδή έχει και θετικές και αρνητικές στοιχές αυτή τη στιγμή. Ακόμα και σε προγράμματα Interreg δηλαδή δεν μπόρεσαν να ενσωματωθούν οι GTC γιατί το Interreg ακριβώς γεννήθηκε για να υποστηρίξει την διασυνοριακή συνεργασία. Και εντούτοις σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα Interreg ή GTC. Έχουν καθοριστεί λοιπόν η GTC ως προτεραιότητα στα πλαίσια της διεθνικής ε, συνεργασίας αλλά οι δυσκολίες δεν έχουν εντοπιστεί μόνο με τα, με Interreg. Έχουμε και προγράμματα Life και Cosme υπό τον εθνικό έλεγχο και στα οποία επίσης δεν μπορούν να συμμετάσχουν οι GTC, το URBACT, στα οποία δεν προβλέπεται η δυνατότητα χρηματοδότησης ε, έργων που προέρχονται από τους ομίλους. Μόνο στο Interact έχουμε θετική συνεργασία, αλλά και εδώ χωρίς άμεση χρηματοδότηση κανένας έργου. Δηλαδή, έχουμε δημιουργήσει ένα μέσο που είναι εξαιρετικά δύσκολο να το χρησιμοποιήσει κανείς. Και αυτό εξηγεί την μερική μόνο επιτυχία που έχει γνωρίσει. Επιπλέον, οι όμιλοι αυτοί έχουν νομικό καθεστώς ε, σε διάφορα κράτη, σε διαφορετικά κράτη, τα οποία κράτη θα πρέπει να προχωρήσουν στις ε, εξαιρέσεις του νομοθετικού τους πλαισίου προκειμένου να επιτρέψουν τις λειτουργίες του EGTC, αλλά αυτή η εξαίρεση δεν γίνεται σχεδόν ποτέ. Δηλαδή υπάρχουν και νομικά εμπόδια όπως σας έλεγα. Προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το νομικό πρόσωπο, αυτή η νομική οντότητα που ονομάζεται GTC στις διάφορες χώρες. Αντίστοιχα δεν έχουν αναπτυχθεί οι επαφές με τις τρίτες χώρες. Έχουμε κάποιες συμφωνίες όπως με Μολδαβία και Ουκρανία που προβλέπουν τη δημιουργία μόνιμων δομών για την διασυνοριακή συνεργασία, όμως αυτές δεν έχουν πάρει τη μορφή GTC αυτές οι συμφωνίες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαγράψουμε το όλον τραβώντας ένα τεράστιο χ από πάνω. Δεν είναι όλα άχρηστα, δεν είναι... Βλέπουμε για παράδειγμα ότι η συμμετοχή αυξάνεται, εγγράφονται όλο και περισσότεροι όμιλοι, η GTC, στο σύνολο, αναπτύσσουν τον προϋπολογισμό τους υλοποιούν τις δραστηριότητες τους, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε μία υποστήριξη στο επίπεδο της επικοινωνίας, της επιφάνειας και στις ε, δυνατότητες ε, έκφρασης ε, και συνεργασίες σε μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Αν θεωρούμε ότι πρέπει η Ευρώπη να κινηθεί προς την κατεύθυνση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τότε οι όμιλοι εδαφικής συνεργασίας είναι κεντρική σημασίας για την υλοποίηση ενός τέτοιου στόχου. Αυτό μαζί με άλλες δομές φυσικά, τις ε, μακροπεριφερειακές στρατηγικές για παράδειγμα, όπου μπορούν να θέσουν ένα πλαίσιο της συνεργασίας πέραν των συνόρων, δηλαδή της Ευρώπης που δεν θα είναι φτιαγμένη μόνο από τα κράτη, αλλά από περιοχές με διαφορετικές περιφέρειες που θα συνεργάζονται μεταξύ τους ώστε να οδηγήσουν εν πάση τόση σε μια πραγματικά πολυεπίπεδη Ευρώπη που θεωρώ ότι χρειαζόμαστε άμεσα. Σας ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Έχουμε έναν εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν, ο κύριος Αλεξάνδερ Φέστελ, αν το λέω καλά, πάλι λέει Πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την ε, έκθεση και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ο EGTC είναι και παραμένει για μας σημαντικό όχημα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, ιδιαίτερα φυσικά για διασυνοριακά προγράμματα. Έχει βοηθήσει και στο παρελθόν και εξακολουθεί να βοηθεί στην υλοποίηση, αλλά βεβαίως προχώρησε κάπως πέραν αυτού και θεματικά Βλέπουμε στα EGTC από νοσοκομεία μέχρι δίκτυα κινητικότητας, όπως και ξεπέρασε το πεδίο εφαρμογής των προγραμμάτων Interreg, που ούτε και αυτό είναι αρνητικό. Σχετικά με την εφαρμογή του νέου κανονισμού, είναι πρόωρο να βγάλουμε συμπεράσματα. Θα υπάρξει η έκθεση της Κομισιόν μέχρι τον Αύγουστο του 2018. Αυτό που μπορούμε να δούμε από τους 56 υφισταμένους GTC είναι ότι ένα εξαιρετικό μέσο που εξασφαλίζει την θεσμική συνεργασία και τον συντονισμό. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η μεταφορά από ad hoc νομικές λύσεις σε σταθερότερες δομές είναι μια πολύ σημαντική διάσταση. Ως προς το μέλλον εμείς θα εξακολουθήσουμε να χρησιμοποιούμε το input και την βοήθεια των NGTC στα πρόγραμματα Interreg και συμφωνούμε και, και ευχαριστούμε και την Επιτροπή των Περιφερειών και το Κοινοβούλιο για την ε, βοήθειά τους στην ε, υποστήριξη των NGTC. Δόκτωρ Σέλμερ, μπορείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις και τα σχόλια ε, ίσως να ευχαριστήσω ιδιαίτερως ε, όλους όσους επένεσαν τη δουλειά μας και μερικά πολύ λίγα σχόλια. Σε ό,τι αφορά το ιστορικό δεν αναφερθήκαμε σε αυτό στην έκθεση γιατί έχουν λεχθεί πολλά παλιότερα, έχουν γραφτεί πολλά, εστιάσαμε πιο πολύ στο μέλλον για να εξάγουμε συμπεράσματα για το τι χρειάζεται να γίνει όπως είπε ο κ. Τσέλερ. Θέλαμε να υπογραμμίσουμε τις δυσκολίες, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Επίσης, αναφέρουμε και συγκεκριμένες θετικές εμπειρίες. Δεν μπορώ να πω ότι το, το ε, εργαλείο αυτό δεν χρησιμοποιείται εξαιτία των δυσκολιών και του Interreg. Εμείς έχουμε δει επιτυχίες σε ορισμένους ομίλους εδαφικής συνεργασίας που ξεπερνούν τη χρήση των πόρων Interreg. Ε, τα πράγματα όμως θέλουν το χρόνο τους. Ε, τα διάφορα ζώα μεγαλώνουν και ενηλικιώνονται με διαφορετικούς ρυθμούς. Έτσι είναι και τα εργαλεία που διαθέτουμε. Αν, θέλουμε, αν θέλετε περισσότερη ολοκλήρωση ε, στις μεθοριακές ζώνες θα πρέπει να έχουμε και υπομονή, να έχετε και υπομονή και χρειάζεται και ε, διάδοση γνώσης, χρειάζεται πειθό, χρειάζεται ε, εκμάθηση, εκπαίδευση. Το σημαντικό είναι να διδασκόμαστε από τι εμπειρίες μα, έτσι ώστε να δούμε ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα προκειμένου να βελτιωθεί το νομικό πλαίσιο των ομίλων αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τσέλερ. Θέλετε το λόγο ξανά. Ένα μικρό σχόλιο. Δεν κατηγορούμε τους υπαλλήλου της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα σχόλια αυτά. Αλλά θα ήθελα να απευθύνω μία έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την έκθεση για τη συνοχή και αν όντω είναι τόσο σημαντική η διασυνοριακή συνεργασία, θα πρέπει να αναφέρεται αυτό στην έκθεση για την συνοχή, να μην το παραβλέπουμε αυτό. Το κοινοβούλιο ήταν αυτό που πρώτο αναφέρθηκε στα μέτρα που, και στα εργαλεία που υπάρχουν για τη διεθνωριακή συνεργασία και νομίζω ότι το ίδιο παράδειγμα θα πρέπει να ακολουθήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε απόλυτο δίκιο, λέει η Πρόεδρος. Το αναφέραμε αυτό στην έκθεσή μα. Και μάλιστα το τονίσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση, για τη μελέτη. Εν συντομία ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια έκθεση για την εφαρμογή, για την υλοποίηση αυτού του εργαλείου κάποια στιγμή. Όποτε είναι θεωρηθεί ε, ε, επίκαιρο. Ναι, καλή ιδέα λέει ο Πρόεδρος. Ας δούμε και τις υπόλοιπες εκθέσεις για την εδαφική συνεργασία και μετά θα μπορούσαμε να εκδώσουμε και μια έκθεση πρωτοβουλία για τους ομίλους εδαφικής συνεργασίας. Ευχαριστούμε. Η Επιτροπή μας επιθυμεί να παρακολουθεί την εξέλιξη διαδικασία, να ενημερώνεται. Και Ας έχουμε στο μυαλό μας ε, ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνοι υπουργοί και θα πρέπει να τους ε, απασχολούμε και να τους ενοχλούμε και για αυτό το ζήτημα, όχι μόνο για το, τα επιχειρησιακά σχέδια. Ωραία. Όσοι είμαστε παρόντες έχουμε την, ε, την τιμή να εγκρίνουμε τις ε, αποφάσεις των συντονιστών η συνάντηση των συντονιστών έλαβε χώρα νωρίτερα σήμερα. Ε, οι αποφάσεις διανεμήθηκαν. Αν δεν έχετε σχόλια... Α, ναι, έχουμε ένα σχόλιο. Ο Βανίστεροι. Είδαμε τα, έχουμε τα πρακτικά όλα πολύ σωστά. Ένα σημείο θέλω να σχολιάσω το 7. Να προσθέσω κάποιες πληροφορίες σχετικά με την ε, κατάσταση σε ό,τι αφορά το ψήφισμα για την απλοποίηση. Ε, ναι, ναι, ωραία. Εκεί αναφέρει τρεις συντονιστές είπαν ότι δεν είχαν αρκετό χρόνο οι ομάδες τους. Θα ήθελα να προσθέσουμε ότι οι φιλελεύθεροι δεν διαφώνησαν. Οι τρεις πρώτοι συμφώνησαν, οι φιλελεύθεροι δεν διαφώνησαν. Μια πολύ μικρή ε, Μπορώ να σας δώσω το κείμενο. Ωραία, ναι, όπως αφηνίζει την κατάσταση. Αν μπορείτε να μας δώσετε γραπτό το κείμενο, πολύ καλά. Περνάμε στα διάφορα. Υπάρχουν άλλα θέματα. Όχι. Να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας θα λάβει χώρα στις 30 Νοεμβρίου το απόγευμα 3 με 6.30 και την 3